Colleagues, we're going to make a prompt start. People uh, need to get away, and I'm conscious that uh, this is a big imposition, having votes this afternoon, so we're going to make a prompt start. Να ξεκινήσουμε λοιπόν συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Στο σημείο 7, 10, 11, 13, 15 αναβλήθηκαν. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στην ατζέντα, εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη κρατικά και Ιρλανδικά δεν θα έχουμε σήμερα. Οι συστάσει των συντονιστών σύμφωνα με τον κανονισμό 205 και για την διοργάνωση επιπρόσθετη συνεδρία στι 9 Μαου στο Στρασβούργο. Συμφωνεί, παρακαλώ, η Επιτροπή μα μάλιστα. Συμφωνεί. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι κανείς που δεν έχει την κάρτα του μαζί. να ξεκινήσουμε στις δύο. Ξεκινάμε. Ε, αν ε, τυχόν έχετε ξεχάσει πουθενά την κάρτα σας, στην Ολομέλεια, πείτε μας για να σας ε, βοηθήσουμε, γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε πάρα αυτά σήμερα, μην καθυστερήσουμε. Κανείς άλλος, γιατί πρέπει να φύγει και πολλοί κόσμοι μετά τις ψηφοφορίε. Κανείς, έτσι. Ωραία. Just checking with coordinators that everyone... Οι συντονιστές παρακαλώ είναι έτοιμοι. Πολύ ωραία. Όλοι έτοιμοι. Σημείο 4. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την εφαρμογή του νόμου σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και την κατάρτιση Europol και έκλεισε των αποφάσεων 2.09.371 και 2.05.681 Αγκουστίν Δία Μέρα. Ο εισηγητής. Ψηφίζουμε. Αγαπητέ εισηγητά, θέλετε να πάρετε το λόγο. Αν όχι, θα ψηφίσουμε πάρα αυτά. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή βρισκόμαστε στο τέλος ε, ενός ε, μιας μακράς διαδρομής. Ε, νομίζω ότι θα ήταν ευγενές εκ μέρους μου να ευχαριστήσω θερμόλες και όλους τους συνεδέλφους και να ευχαριστήσω όλους ιδιαιτέρως τους Γκάι, Αντουάν και εσάς προσωπικά. Κύριε Διαδεμέρα, συγγνώμη, αλλά κάποιο πρόβλημα έχουμε τεχνικό με την διερμηνία. Αν θα μπορούσατε παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τι πρόβλημα υπάρχει. Okay, have another go, Mr. Diaz de Mera. Please, uh, if you can repeat what you said όταν τα επαναλάβετε αυτά που είπατε κύριε Εντή Ναι, είναι πολύ εύκολο να πω αυτά που είπα. Είπα ένα θερμό ευχαριστώ, ευχαριστώ από καρδιά σε όλους τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους από τις πολιτικές ομάδες που συμμετείχαν και ακολούθησαν αυτή τη μακρά διαδρομή που ολοκληρώνεται. Και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τώρα τον Αντουάν και εσάς προσωπικά. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Δίας. Θα μέρα πάμε πάρα αυτά στην τροπολογία 3. Έναρξη παρακαλώ ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. Και έτσι περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία λέω. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 40 ψήφοι υπέρ 3 κατά 2 αποχές. Συγχαρητήρια αγαπητέ Ισίδα. Στο 5 περνάμε σε ό,τι αφορά τι συνθήκε εισόδου και κατοικία επικών τριτών χωρών σε ό,τι αφορά την έρευνα με ε, και το καθεξής ε, Μετά από την παρουσίαση του σχεδίου α, ε, της οδηγίας για τους ε, σπουδαστές και τους ερευνητές της 11 Απριλίου, δεν έχουν καταβληθεί ε, τροπολογίες και γι' αυτό λοιπόν σύμφωνα με τον ε, κανόνα 66, άρθρο 66 θα περάσουμε στην ε, ψήφιση του σχεδίου συστάσεων. Δεν είναι εδώ η κυρία Βίξτρομ. Ψηφίζουμε λοιπόν πάρα αυτά. Έναξη ψηφοφορίας. The vote is closed. And that is carried 40 votes. Εγκρίθηκε 40 ψήφοι υπέρ, 5 κατά μία εποχή. Ε, συγχαρητήρια στην ε, εισηγήτρια και στο γραφείο της. Συνάδελφοι, πάμε στο 6. Καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων σε εξωτερικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Μποντήλ Βαλέρο, η συγγήτρια. Αν δεν θέλει το λόγο, θέλει. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω το λόγο για να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ λοιπόν που βοηθήσατε για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Αυτό ήθελα ουσιαστικά να τονίσω, την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Ε, περνάμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συμβαστική 1. Ε, έναξη. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 2. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 16 παρακαλώ, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η 17. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η 18. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τρία Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 3. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Ε, Τροπολογία 25. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Συγγνώμη. 25 δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, με ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίθηκε. 27. Πέρας. Εγκρίθηκε. 28 ψηφίσμα. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 9 ψηφίσμα. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 33. Ψηφίζουμε. Πέρας. Η 35. Εγκρίθηκε. 35 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 1α ψηφίζουμε. Πέρας. Εκρίθηκε. Η συμβαστική 4α. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εκρίθηκε. Συμβαστική 10. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 5. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 43. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 44. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 45. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. Η 46. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. 47 πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 48 ξεχωριστή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 49. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 56. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκριθήκε η 57. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 60. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η 63. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 66. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 64. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 65. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 68. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 71. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 72 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίθηκε. 74. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 75 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 76 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορριφθήκε. 77 σε τμήματα. Έχει αιτηθεί σοσιαλιστές και δημοκράτες. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Α, όχι, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, πάμε κατευθείαν στο δεύτερο τμήμα. Στο δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Όχι, στο πρώτο τμήμα. Πολύ να με συγχωράτε, στο πρώτο τμήμα ψηφίζουμε, Τη 77. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει με αυτή την τροπολογία, λέει ο Πρόεδρος. Στο δεύτερο τμήμα, λοιπόν, ας ψηφίσουμε. 79. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε 80. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε 86. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 87. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. 99. 80 είναι, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 91. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκριθήκε. 92. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 93. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. 94 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκριθήκε. Και πάμε στις λογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε η τρία. Πέρας. Εγκρίθηκε η τέσσερα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε η πέντε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε η 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε η 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε η εννέα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Επί του συνόλου του κειμένου τώρα ψηφίζουμε παρακαλώ. Έναρξη έκτακτης ψηφορίας. Πέρας εγκρίθηκε 46 ψήφοι υπέρ, 0 ψήφοι κατά και 5 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Βαλέρο, την εισηγητρία. Colleagues, now we move to point 8. Περνάμε στο 8 τώρα. Προσωρινά μέτρα για την διεθνή προστασία προ όφελο τη Σουηδία βάσει του άρθρου 9 τη απόφαση 2015-1523 του Συμβουλίου και του άρθρου 9 της απόφασης του Συμβουλίου 2015-1601 στο για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Σκακέλερ είναι η συγγήτρια. Προτείνει η συγγήτρια να απορρίψουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με το 17 02 θα ψηφίσουμε πρώτα την ε, πρόταση της εισηγητρίας να απορριφθεί το κείμενο της Κομισιόν και αν ε, υπερψηφιστεί αυτή η πρόταση θα ψηφίσουμε μόνο την τροπολογία στην την πρόταση της ε, θα ψηφίσουμε δηλαδή τις τροπολογίες της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά το σύνολο και τέλος το σύνολο του κειμένου και τέλος το νομοθετικό κείμενο να ρωτήσω την κυρία Σκάκελη αν θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Πολύ ωραία. Α, πάμε να ψηφίσουμε λοιπόν. Αν ε, θέλετε το λόγο, μην διστάσετε να το ρωτήσετε. Ας ψηφίσουμε. Ονομαστική κλίση, προφανώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. here. So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 23 προς 30. Amendment 8. The vote is open. Η τροπολογία 8 άρχεται τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 4. Γράφεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5. Έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 6. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 7. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε αρχή ψηφοφορία. Περιμένω το συντονιστή μου να μου πει τι, θα, κάνω, τι να κάνω. Και τώρα, η τροπολογία 2 το νομοθετικού ψηφίσματος, η ψηφοφορία. Είναι τροπολογία 2, έτσι δεν είναι. Τροπολογία 2. Ψηφίσατε όλοι. Καταλάβατε όλοι τι πρέπει να ψηφίσετε. Συμφωνήσατε. Ωραία. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Εδώ και ώρα δηλαδή έχει αρχίσει. Πέρας. Απορρίπτεται. 37 κατά 14 υπέρ. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. vote is closed. Εγκρίθηκε 27-23 και μία αποχή. Thank you to the rapporteur. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Colleagues, we move to our final vote. Πάμε στην τελευταία μας ψηφοφορία. Η παγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας ΤΑΔΕ κτλ. σε μέτρα ελέγχου. Η συγκητής είναι ο κύριο Μπόνι. Δεν ξέρω, θέλετε το λόγο κύριε Μπόνι. Θέλετε το λόγο πριν ψηφίσουμε. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν, χωρίς τροπολογίες. Είναι μία και τελική ψηφοφορία ίδια, αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 51-0 με μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Μπόνιο. Λοιπόν, συνάδελφοι, πάμε αμέσω στα υπόλοιπα της μέσης διάταξης. διάταξη. θα συνεχιστεί αμέσω η συνεδρίαση. So, let's... Η κυρία Γκόμες προεδρεύει. Επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση. Με χαρά καλωσορίζω την Επίτροπο κυρία Γιούροβα. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε μαζί της. The umbrella agreement and Την Ελλάδα και άλλα θέματα ε, που μας ενδιαφέρουν. Πώς θα το ε, οργανώσουμε πρακτικά. Θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο πρώτα για να ακούσουμε την παρουσίαση. Ε, το θέμα είναι όχι, όχι Ελλάδα, το ΕΚΡΙΣ, το ΕΠΟ και άλλα τέτοια θέματα. Ε, θα κάνουμε ερωτήσεις στη συνέχεια συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων και θα έχει χρόνο για να απαντήσει η Επίτροπος. Και θα υπάρξει και δεύτερος γύρος ερωτήσεων, ε, όσα μέλη θέλουν να ρωτήσουν και μετά να απαντήσετε εσείς κυρία Επίτροπε. Θα πρότεινα οι βουλευτέ που θα πάρουν το λόγο να προσπαθήσουν να περιστούν σε ένα δίλεπτο έταστος Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσουμε αμέσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Γιούροβα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συνεχίσω μαζί σας ε, το διάλογο και κυρίως ε, σήμερα θα ασχοληθώ με το ποινικό, ε, την ποινική δικαιοσύνη. Μετά τον τελευταίο Διαρθρωμένο ε, διάλογο του Οκτωβρίου του 2015 βίωσε η Ευρώπη τρομερές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανέωσε και ενίσχυσε τις πρωτοβουλίες της ε, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις αρχές μας. Ε, η δικαστική συνεργασία στα ποινικά θέματα είναι ένα μέρος της απάντησης και με αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το υπόβαθρο, έχουμε προτείνει μια τροποποίηση του έγκρις για την καλύτερη ανταλλαγή ε, πληροφοριών ε, σε σχέση με το ποινικό μητρό υπηκών τρίτων χωρών. Χαίρομαι που βλέπω ότι ο συγητής κύριος Κέρκοπ ξεκίνησε ήδη να εργάζεται πάνω σε αυτή την πολύ σημαντική πρόταση η οποία πιστεύω θα βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα επίσης να σας προειδοποιήσω ε, για την επόμενη συζήτηση που θα γίνει σε επίπεδο Υπουργών Δικαιοσύνη και στο Άμστερνταμ ε, το Γενάρη ε, εσείς είχατε κύριε Πρόεδρε Μωράης α δεν είναι εδώ ο κύριος Μωράης τέλος πάντων ελπίζω να με ακούει είχε ε, παραστεί πάντως και αυτό ήταν η αφετηρία η Ολλανδική Προεδρία θέλει να προωθεί συστήματα συνδρομής σε κάποιες χώρες αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να δούμε ποια είναι τα όρια και αν αυτά ε, είναι επαρκή απέναντι στην ψηφιακή εποχή. Γιατί μιλάμε για την λεγόμενη ψηφιοποίηση του ποινικού δικαίου. Προτείνουμε και στοχευμένε τροποποιήσει στην οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο, διότι είδαμε ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Θα εξετάσουμε το πώς μπορούμε ε, να βελτιώσουμε τη δράση των μονάδων ε, ανταλλαγής ε, πληροφοριών, fuse όπως λέγονται, και θα δούμε τι γίνεται με τις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες για να είναι πιο ασφαλής χωρίς να απαγορευτεί ταυτόχρονα και αυτό το πολύ σημαντικό μέσο πληρωμής. Μετά την κρίση με τα έγγραφα του Παναμά επανέρχεται και το ζήτημα της διαφάνειας, το οποίο εσείς και ιδιαίτερα η συγκίτρια κ. Σατζεντίνη έχετε ήδη τονίσει ε, στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων. Στόχος μου είναι να σας παρουσιάσω μια αναθεωρημένη πρόταση τον Ιούνιο. Πέραν λοιπόν των προληπτικών αυτών μέτρων έχουμε να προτείνουμε μέχρι τα τέλη του έτους ε, και την αμοιβαία αναγνώριση της ε, λήψης απόφασης για, την, για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων ε, όταν λαμβάνεται η απόφαση αυτή από το δικαστή μιας χώρας να αναγνωρίζεται από τις κασίε αρχές των άλλων κρατών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, είμαι περήφανη διότι ολοκληρώσαμε τη μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων και θέλω ε, να αποτίσω φόρο τιμής στον εισηγητή Άλμπρεχτ ε, και στην κυρία Λοριστίν για τη δουλειά τους. Από κοινού πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα άρτιο μακρόπνο αποτέλεσμα. Και τώρα θα εστιάσουμε στην αποτελεσματική υλοποίηση ε, των σχετικών διατάξεων ε, από τα κράτη-μέλη, ώστε όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις ε, να ωφεληθούν από αυτό το Big, Bang, την έναρξη ισχύω δηλαδή του κανονισμού αυτού. το 18 συγκεκριμένα την Άνοιξη προβλέπεται η ισχύ και έτσι θα δώσουμε τα σωστά μηνύματα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα στηρίξουμε όμως και τις επιχειρήσεις και την καινοτομία στην ψηφιακή ιστορική εποχή. Επίσης θα εστιάσουμε την αμοιβαία και την αποτελεσματική συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου με τη σχετική οδηγία. Χρειαζόμαστε να υπάρξει αναβαθμισμένη προστασία και κατά την ε, μεταβίβαση δεδομένων ε, ένθεκα και του Ατλαντικού. Αύριο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την υπογραφή της Γενικής Συμφωνίας ε, που θα θεσπίζει ένα ισχυρό πλαίσιο και κανόνες για την προστασία δεδομένων, για την ε, διμερείς διακανονισμούς ε, της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας που ισχύουν μεταξύ της Ένωσης των κρατών μελών της και των ΗΠΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα προσωπικών δεδομένων στον τομέα των εμπορικών ε, συναλλαγών, Θέλουμε οι συστάσεις που διατύπωσε η ομάδα εργασίας του Άντρου 29 να εφαρμοστούν. Επίσης προχωρήσαμε και σε ό,τι αφορά το πακέτο των δικαιωμάτων σε περίπτωση της ε, ε, πολιτικής δικονομίας, διαδικαστικά δικαιώματα. Ο κ. Ντεγιόγκ έχει την πλήρη υποστήριξή μας για να καταλήξει σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα και σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, το εύρος. Τώρα γιατί ειδική κατάσταση των παιδιών προσφύγων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πάντοτε ε, πρώτο μου μέλημα είναι η, είναι η αντιμετώπιση των αναγκών τους, είτε στα hot spot, είτε αν για συνόδευτα παιδιά η φροντίδα τους, είτε ε, η ένταξή τους ε, στην κοινωνία πρέπει να πετύχουμε, πρέπει να φέρουμε σε πέρα ε, το καθήκον Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ε, τι έχουμε κάνει για την ε, αντιμετώπιση της παρότρινσης σε μίσος. Ε, θέλουμε έναν κώδικα διοντολογίας μέχρι τον Ιούνιο. Η ελευθερία λόγου πάντοτε βέβαια είναι σεβαστή, όμως πρέπει το ίντερνετ να μην είναι ένας χώρος ε, χωρίς νόμο, ε, εκτός νόμου. Με τις ποινικέ αρχές θέλουμε επίσης ε, να ολοκληρώσουμε και τη διαδικασία για την σύσταση του, Ευρωπαϊκού, του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Στόχος είναι να έχουμε ολοκληρώσει εντός του έτους. Η Ολλανδική Προεδρία δείχνει δεσμευμένη να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτό και την ευχαριστώ για αυτό και με τη Σλοβακική Προεδρία στην Βρατισλάβα θα έχω αύριο συζητήσει επ' αυτού. Νομίζω ότι κάνουμε σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο σε αφορά ε, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα κράτη-μέλη θεωρητικά στηρίζουν τα βασικά ε, σημεία της πρότασης, επί τη βάση όμως του ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα. Τώρα λοιπόν ολοκληρώνουμε την πρώτη ανάγνωση των ε, εναπομεινών των κεφαλαίων. Η θέση μου στις διαπραγματεύσεις πάντα ήταν και παραμένει ότι πρέπει να έχουμε ένα ανεξάρτητο και αποτελεσματικό γραφείο ε, Ευρωπαίου Αγγελέα. Και θα πρέπει να ξεκάθαρες ε, οι αρμοδιότητες και σαφής ε, η προτεραιότητα. Είναι σαφής ε, η επιχειρηματολογία μας και επιβεβαιώνεται και από το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών και πρέπει να την τηρήσουμε. Οι διατάξεις ε, για τις επικουρικές αρμοδιότητες θα πρέπει να είναι εξισορροπημένες για να μην στερηθούν, για, για να μην στερηθεί κάποιον αρμοδιοτήτων ε, το γραφείο αυτό από, το, την πίσω πόρτα. Δεύτερον, το Συμβούλιο άλλαξε σημαντικά την παλιά δομή που προτινόταν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επιθυμεί το Συμβούλιο να λειτουργεί ως συλλογικό σώμα η Εισαγγελία. Και πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι Υπάρχει, και εθνικός σύνδεσμος στην εισαγγελία και επιμένει οι Ευρωπαίοι ε, εισαγγελείς να επιβλέπουν ε, τις περιπτώσεις και να αποπτεύουν τις υποθέσεις στα κράτη-μέλη. Άρα θα ε, πρέπει να δημιουργηθούν μόνιμα τμήματα εισαγγελίας που θα μπορούν να εκχωρούν αρμοδιότητα σε εισαγγελείς των κρατών μελών να εξετάζουν και να χειρίζονται υποθέσεις. Αλλά αν είναι υπερβολική χώρηση αρμοδιοτήτων, τότε αμφισβητείται η ίδια ύπαρξη των τμήματων της εισαγγελία των μονίμων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εκχωρείται η αρμοδιότητα από τον ένα ευρωπαϊκό σε, μάλλον εισαγγελέα σε άλλο, ε, και η υπερβολική χώρηση να περιορίζεται σε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις για να μπορεί να έχει ένα εποπτικό ρόλο και να ασκεί ε, αρμοδιότητες και να είναι ουσιαστική η πολιτική μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ελπίζω επίσης να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, στον κανονισμό του Eurojust για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και να βελτιώσουμε την λειτουργία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν καλύτερα τη Eurojust, ιδιαίτερα ε, τις κοινέ ομάδες έρευνας και δίωξης ε, που υποστηρίζουν ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πρέπει να καλύπτουμε τα κενά, να προτείνουμε βελτιώσεις και να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην εφαρμογή και στην επιβολή, ε, έτσι ώστε όλη αυτή η νομοθεσία να γίνει πραγματικότητα στην πράξη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το κεκτημένο μας δεν ε, έχει απορροφηθεί από τα κράτη-μέλη. Ε, η μεταφορά δεν είναι πάντα ενιαία, πολλές φορές είναι εμβαλωματική και άσχετα θέματα μεταξύ τους θα πρέπει οι δικαστές και οι εισαγγελείς ε, παντού στην Ευρώπη να εφαρμόζουν ε, με τον ίδιο τρόπο το ποινικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό, για να δημιουργηθεί μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μόνο έτσι θα λειτουργεί ο χώρος της δικαιοσύνης με εκτελεστικά μέτρα και μέτρα δίωξης και έρευνας διασυνοριακά συνεχίζονται οι ταυτόχρονες κοινέ προσπάθειες τρομοκρατικών δυνάμεων ε, των σωμάτων ασφαλείας σε διάφορα ε, Είναι καλή, αλλά έχουν γίνει και λάθη και καθυστερήσεις υπάρχουν. Θα πρέπει να εφαρμόζονται σωστά όλα τα μέτρα και λιμένες αποφάσεις. Αυτό τι σημαίνει. Από τη μια πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των προτέρων να βοηθάει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ε, τα κεκτημένα, τα εγχειρίδια, τους εμπειρογνώμονες και να ε, κάνει σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ε, δεν θα πρέπει όμως να ε, δείχνει ατολμία σε περίπτωση προσφυγής επί να προσφέρει όταν υπάρχουν παραλήψεις ή παραβάσεις για να καταπολεμώνται οι ολιγορίες. Το Μάρτιο στο Συμβούλιο συζητήσαμε ε, τα θέματα αυτά και μετά τη διάσκεψη που ε, διοργάνωσα για τη ριζοσπαστικοποίηση ε, τον Οκτώβριο, ιδιαίτερα για τη ριζοσπαστικοποίηση των κρατουμένων στις φυλακές. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν σε αυτή. Και μεταξύ αυτών είναι οι ελληνές συνθήκες που επικρατούν σε κάποιες ευρωπαϊκές φυλακές. σε ένα γράμμα που έστειλα, εξήγησα όλα αυτά τα θέματα και πρότεινα κάποιες λύσεις. Επίσης, εξήγηλα ε, τη σύσταση ομάδας ε, υψηλού επίπεδου που βάσει των συστάσεων θα προχωρήσει, που κάνει η υποομάδα για τα σοφρονιστικά καταστήματα, να ανταλλάσσουμε ε, βέλτιστες πρακτικές, οι χώρες που θίγονται περισσότερο και είμαι σε επαφή με τον πρόεδρό σα. Σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή σα για τα θέματα αυτά, υπό την αιγίδα της κυρίας Ινετβέλτ. Τα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον μαζί με τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμανς. Η λειτουργία ε, των δικαστικών συστημάτων είναι σημαντικό τμήμα του κρατούς δικαίου και επιτρέψτε μου ε, επευκαιρία να σας ενημερώσω για τα βασικά συμπεράσματα της τέταρτης προσθήκης ε, που δημοσιεύσαμε στον πίνακα επιδόσεων το scoreboard. Ξέρετε ότι αυτό βοηθάει τα 28 κράτη-μέλη για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, την ανεξαρτησία της και τη λειτουργία της. Έχουμε συγκριτική ενημέρωση, αυτά τα τρία στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη. Γενικά, τα περισσότερα κράτη-μέλη προοδεύουν για να βελτιώνουν τα συστήματά τους, τα δικαστικά και ε, Υπάρχουν και κάποια σεθαρρυντικές τάσεις από την πρώτη φορά που είχαμε δημοσιεύσει αυτό το πίνακα. Αυτό φορά αστικές, εμπορικές υποθέσεις, υπάρχει βελτίωση εκεί, ωστόσο στο διοικητικό στα διοικητικά δικαστήρια έχει επιδεινωθεί και η ποιότητα. Μπορεί να βελτιώνεται ε, η μηχανοργάνωση ε, σε ό,τι αφορά διαδικασίες επιγραμμικές για μικρές αξιώσεις, αλλά χρειάζονται και άλλες προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάρτιση των δικαστικών και να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και για τις διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Ο πίνακας επιδόσεων, το scoreboard, είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται και φέτος για πρώτη φορά περιλαμβάνει και έρευνες του Ευρωβαρομέρτου για την ε, αίσθηση που έχει ο κόσμος για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των δικαστηρίων. Και εδώ μιλώ για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Λένε λοιπόν οι χρήστες ότι διαφέρει η κατάσταση από κράτος σε κράτος. Υπάρχουν χώρες όπου είναι χαμηλή η αντίληψη για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης διότι υπάρχουν πιέσεις ή επεμβάσεις από πλευράς της πολιτικής ή της κυβέρνησης, οικονομικών και άλλων συμφερόντων και η δικαιοσύνη δεν είναι απολύτως ανεξάρτητη. Αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και παρακολούθηση. Αξιότιμα μέλη, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, κάλυψα εν μέρη μόνο τα θέματα τα οποία ε, είναι του χαρτοφυλακίου μου και περιμένω με χαρά να ακούσω τις ερωτήσεις σας για να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε αμέσως με τους συντονιστές. Κύριε Χολμάιερ, δεν είναι εδώ νομίζω. Ο κύριος Μπόνι θα μιλήσει εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Επίτροπε, και μεγάλη χαρά που σας ξαναβλέπουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης ε, και για την επιστολή, την επεξηγητική για τα ζητήματα αυτά. Είναι σημαντικό το ότι είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τα κάποια θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έχω κάποια σημεία να επισημάνω. Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ περισσότερο με... και για την ανταλλαγή πληροφοριών και στο πλαίσιο του έκρης. Είναι απαραίτητο, το χρειαζόμαστε. Και οι προτάσει σας για την χρήση ψηφιακών εργαλείων στον τομέα του ποινικού δικαίου και σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ και Και νομίζω ότι θα καταστήσουν ε, πολύ πιο γρήγορε πολλέ από τι διαδικασίε αυτέ. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραφεί μια συμφωνία γενική πλαίσιο, όπως αναφέρεται αύριο. Ε, υπάρχουν κάποιε ερωτήσει από την πλευρά τη Επιτροπή, Λίμπε, αλλά θα πρέπει να σα υποστηρίξουμε. Σα ευχαριστώ επίση για τη συνεργασία σα με όλου του εταίρου και κυρίω ε, σε ό,τι αφορά την ομάδα του άρθρου 29 σε ό,τι αφορά την ασπίδα προσωπικών δεδομένων. Και είμαι βέβαιος ότι σε τελική ανάλυση θα καταλήξουμε στην ε, πιο ενδεδειγμένη λύση. Σημαντικό είναι επίση αυτό που είπατε για τι ομιλίες που ε, οθούν στο μίσος και θα υπάρξει και ένα κώδικα θετολογίας και το δικό σας το έργο, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή με τους παροχούς διαδικτύου θα ολοκληρωθεί ακριβώς με τον κώδικα τεντολογίας αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί είναι σημαντικό φυσικά να υπάρχει ασφάλεια, να υπάρχει συγγνώμη, ελευθερία στο διαδίκτυο αλλά χρειαζόμαστε παράλληλα και κάποια εργαλεία για να πατάξουμε ορισμένες μορφές όπως για παράδειγμα οι ομιλίες μίσους. Να σας ρωτήσω επίσης ε, τα περαιτέρω βήματα για την προστασία των δεδομένων με το GPS και τη σχετική οδηγία δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η δουλειά. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο εφαρμογής ιδιαίτερα για το GPDR που περιλαμβάνει πολλά μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ευελιξία που μεν χρειάζεται δεν θα μας οδηγήσει από την άλλη σε 28 διαφορετικά προγράμματα και συστήματα. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αντιμετωπίσει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ, λέει η κυρία Σύπολη, σε δύο-τρία ζητήματα, έχοντας υπόψη ότι και οι άλλοι συνάδελφοι ενδεχομένω να θέσουν επιπλέον ερωτήματα σε ό,τι αφορά την ασπίδα προσωπική ε, σφαίρα. Πολλέ είναι ανησυχίε. Δύο με αναφέρω δεκτικά. Η κυβέρνηση τη Αμερική δεν ε, αποκλεί την μαζική ε, συλλογή δεδομένων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το αποκλεί τελείω το ενδεχόμενο. Πώ ε, συμβαδίζει αυτό με την ευρωπαϊκή αξία ότι η μαζική συλλογή δεδομένων δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται αναλογική και ενδεδειγμένη ω μέτρο. Και επίσης είναι ανακύπτει πάντα το θέμα του κατά πόσον έχει επαρκείς αρμοδιότητες το άτομο για να ενεργήσει ή κατά πόσον όντως ε, υπάρχουν μηχανισμοί και συστήματα ένδικης ε, καταγγελίας. Αν θα θέλετε να μας απαντήσετε. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την Γενική Συμφωνία, τη Συμφωνία Πλαίσιο, ξέρουμε ότι και η Συμφωνία PNR με τη ΣΥΠΑ και το TFTP δεν, δεν καλύπτονται από το Privacy Act της Αμερικής. Η συμφωνία πλαίσιο όμως θα προϋπέθεται ότι θα ίσχυε από αυτή της νομοθεσίας. Πώς ε, εξηγείται λοιπόν αυτή την αντέφαση. Επίσης, ε, το θέμα των ενδικών μέσων ε, συνδέεται με τη ροή των εμπορικών μέτρων. Και φαίνεται δηλαδή ότι εξαρτάται ε, η δυνατότητα ε, χρήση αντικών μέσων από το κατά πόσο θα συμφωνήσουμε με το Privacy Shield. Και τέλο. ότι εδώ το OPPO υπάρχει μία άποψη του Κοινοβουλίου για την εισαγγελία και κατά τη γνώμη σας, πείτε μας, οι θέσει του Κοινοβουλίου σε τι βαθμό λαμβάνονται υπόψη στι τρέχουσε συζητήσει του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ από το ECR ο επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ, Επιτροπέ, και σα ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Δυστυχώ, ο κύριος Κύρκοπ δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα. Έχει ανελημμένε υποχρεώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα ήθελα να κάνει τα παρακάτω σχόλια. Η καταπολέμηση τη εγκληματικότητα και τη τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατή μόνο εφόσον τα κράτη-μέλη αντιδρούν γρήγορα και συνεργάζονται με αποτελεσματικότητα η συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου τα μεμονωμένα ποινικά συστήματα να συνεργάζονται είναι ουσιώδου σημασία αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντο. Η ομάδα του ECR δεν πιστεύει ότι ένα απόλυτα εναρμονισμένο ποινικό σύστημα ή ένα απόλυτα κεντρικό σύστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί αυτό. Η σωστή δέσμευση για την ανταλλαγή χρήσιμων και ωφέλιμων πληροφοριών είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο να πετύχουμε αποτελέσματα. Και ω εισηγητή για τον κανονισμό έκρι, ο κ. Κύρχο προσβλέπει στη συνεργασία μαζί σα και πιστεύει ότι οι τροποποιήσεις που γίνονται σε ό,τι αφορά του υπηκόου τρίτων χωρών είναι ε, απολύτως απαραίτητες. Αυτό έχει να κάνει με την ε, εξίσωση στο ποινικό μας ε, δίκαιο, στις, ποινικά μας συστήματα των ε, τρίτων, τοπικών τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων υπηκών. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτό για να υπάρχει ε, εμπιστοσύνη στην ελευθερία τη μετακίνηση και στην εσωτερική μα ασφάλεια. Θα ήθελα Ευρωπαϊκή... ο κ. Κέρκου να ευχαριστήσει την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπει σημαντική συνεργασία μαζί σα για ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να πλήξουμε του ε, εγκληματίε εκεί που του πονάει, στο πορτοφόλι του, Θα μπορούσε η Επιτροπή να μα πει πώς η Επιτροπή με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος θα βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, ποινικών αρχών για την καταπολέμηση του εγκλήματο όχι μόνο στο πλαίσιο του ΕΠΟ αλλά και σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ανθρώπων και την ε, τρομοκρατία. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις αρχές επιβολής του νόμου να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπος σκοπεύει να κάνει μια αναθεώρηση των κοινών ερευνητικών ομάδων που πάντα τις υποστηρίζει ο κ. Κέρκοπ για να δούμε πώς αυτό το α, πραγματικά α, ωφέλιμο εργαλείο μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Γκρισμπέκ, εξ ονόματο των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω, κυρία Επίτροπε, και να χαιρετήσω ε, τη δέσμευσή σα ε, είναι πραγματικά ε, πολύ ε, αξιόλογη και πολλά τα θέματα και κυρίως ε, περίπλοκα και στρατηγικά όλα. Για αλλαγή, μερικά σχόλια, θα ξεκινήσω από τους βασικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα όταν μιλήσατε για την καταστροφή και ολέθρια κατάσταση που ζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι χιλιάδες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γενικότερα τα παιδιά των μεταναστών ε, φύστανται πολλά δεινά. Έχουμε ένα πρόγραμμα για τα δικαιώματα των ανηλίκων που έληξε, εξέπνευσε, είχε διάρκεια από το 2011 μέχρι το 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα σας ή τη δική σας όθηση έχει σχέδια να φέρει μια νέα πρόταση αποτελεσματική, φιλόδοξη, ε, συνολική με συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προστασία των ανηλίκων και των δικαιωμάτων τους. Δεύτερη ερώτηση. Αυτό που πολύ ωραία αναφέρατε και υπάρχει συνάδελφοι, ε, η γενική συμφωνία και η παρουσίαση της και γενικά η μεταφορά δεδομένων και η μεταβίβασή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εκτός από τη γενική λοιπόν συμφωνία υπάρχει και το Privacy Shield, αλλά θα μπορούσατε να μας δώσετε εσείς περισσότερα στοιχεία και διαβεβαιώσεις ότι ε, η υλοποίηση των δύο αυτών συμφωνιών θα γίνει σε πλήρη αρμονία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Ε, συμφωνία που πολύ πρόσφατα εγκρίναμε στην Ολομέλεια. Θα συμφωνείτε φαντάζομαι. Δεν θα επανέλθω στο άρθρο 29. Ακούστηκε δύο λόγια μόνο πρόεδρε για ε, την εισαγγελία και τον Ευρωπαίο εισαγγελέα. Η αρχική πρόταση ήταν μια κεντρική δομή αρκετά ευρωπαϊκή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αυτό άλλαξε πάρα πολύ, αναθεωρήθηκε 100 ppm των κρατών μελών και είναι πάρα πολύ αποκεντρωμένη η δομή αυτή, πάρα πολύ διακυβερνητική, ε, με ε, εισαγγελείς ε, στους οποίους θα χωρούνται αρμοδιότητες που τους ονομάζεται και συλλογικό σώμα, κολέγιο δηλαδή, αλλά καμία σχέση δεν έχει με την αρχική πρόταση και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρχεντίνη, από των Πρασίνων. Thank Ευχαριστώ. Θα ήθελα να, πω καταρχάς ότι προσβλέπω στην ε, προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την οδηγία, την εθόρυση τη οδηγία για το εξέπλυμα του χρήματο. Χαίρομαι που είπατε ότι δεν εξετάζεται μόνο το θέμα τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, αλλά λαμβάνεται υπόψη και το θέμα των γράφων του Παναμά και εξετάζεται και τα τραστ, τα αυτό θα είναι κάτι ευπρόσδεκτο και ξέρω ότι στο Κοινοβούλιο δεν καταφέραμε να το περάσουμε αυτό και κυρίω λόγω τη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι η πολιτική κατάσταση ενδεχομένω να έχει αλλάξει κάπω στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό να μα επιτρέψει να είμαστε λίγο πιο έντονοι στη διατύπωση σε ό,τι δράσει. Τώρα, για το privacy shield, την αυτή τη προσωπική ε, ζωή. Βλέπουμε ότι οι αρχέ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι το Privacy Shield δεν προστατεύει επαρκώ τα προσωπικά μα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει και το έχουμε θέσει και πολλέ φορέ. Θα ξαναδιαπραγματευτείτε ή τουλάχιστον θα βάλετε μία ρήτρα εκπνοή στην σχετική απόφαση για τη συμφωνία πλαίσιο. Αύριο, από ό,τι κατάλαβα, θα την υπογράψετε. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών αποδέχθηκε τα δεδομένα των επιβατών από το US Privacy Act. Αυτό, ναι, με συγχωρείτε κιόλα, αλλά θεωρώ ότι μειώνει την αξία της συμφωνίας πλαίσιο. Θα ζητήσετε λοιπόν εξαίρεση προτού υπογραφή η συμφωνία πλαίσιο. Και τελευταία ερώτηση για το έκρης, ιδιαίτερα για το άρθρο 4α της πρότασης. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι βάσει δεδομένων που προ... περιέχει εκλη... δεδομένα σε... ότι αφορά εγκλήματα των πολιτών θα περιλαμβάνει και ε, τα στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών με διπλή υπηκότητα. Αυτό δεν αποτελεί διακριτική μεταχείριση και πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει ως διακριτική μεταχείριση τέτοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίτροπε, λέει η Πρόεδρος, θα θέλετε να απαντήσετε μέχρι εδώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Για να βρω τις σημειώσεις μου. How, how I got the, the questions. On, uh, yeah, Mr. several comments on, on... Για το έκρης που είναι ε, τμήμα του θεματολογίου για την ασφάλεια και πολύ σωστά. Γιατί αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υπηκών τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί από τα δικαστήρια. Χαίρομαι για τη θετική ανταπόκριση που λάβαμε όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά και από το Κοινοβούλιο, διότι όλοι αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, φοβόμουν ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα με τη συμπερίληψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Παρόλα αυτά αποφάσισα να υποβάλω την πρόταση με αυτή την μεγιστοποιημένη απέτηση για τη συμπερίληψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, διότι θέλουμε να έχουμε μια ενιαία διαδικασία ταυτοποίησης και βέβαια στο σύστημα αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε και να ε, περιφρουρήσουμε όλα τα ε, πρότυπα για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και καμία παραβίαση της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει επίσης να επεξεργαστούμε την περαιτέρω και το έγκριση αλλά και άλλα συστήματα τα οποία βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου στη διασυνοριακή τους δράση. Έχουμε το Σέγγεν, που προσφέρει φανταστικές ευκαιρίες και είναι θετικό για όλους μας, όμως ε, δίνει και στους εγκληματίες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν ε, και να διαπράξουν αξιόπινες πράξεις όπου πάνε. Άρα δεν έχει σύνορα ούτε το έγκλημα. Γι' αυτό και στο θεματολόγιο ασφάλειας και ποινικής δικαιοσύνης. Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε το δυναμικό της δικαστικής συνεργασίας και των αρχών επιβολής του νόμου, δισαγγελέων, αστυνομίας, για να μπορούν να δρουν αμελητή. Γιατί όλες αυτές οι επιθέσεις που βιώσαμε στην Ευρώπη κατέδειξαν ότι η γρήγορη δράση έχει να σημασία για τη δίωξη των εγκληματίων σε ό,τι αφορά το λόγο μίσους, που, το λόγο δηλαδή που παροτρύνει στο μίσος. Το εντάσσω στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Νομίζω ότι συνειδητοποιούμε ότι δύο τρόποι ριζοσπαστικοποίηση υπάρχουν. Στις φυλακές και στο ίντερνετ. Για το ίντερνετ βλέπουμε ότι κάποιοι κύκλοι, κάποιοι, κάποιες ομάδες ανθρώπων επιθυμούν και θα τα πω μα. Θέλω να ξεκινήσω έναν εμφύλιο πόλεμο στην Ευρώπη. online κάπως ε, βλέπουμε να πραγματώνεται αυτό. Αν διαβάσει κανείς τις συζητήσεις και δει όλα ε, τη ρητορική μίσους. Ήδη υπάρχει δηλαδή αυτό το είδος του εμφύλιος πόλεμο στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα το ίντερνετ είναι και ο τόπος που πρέπει εκεί ακόμα περισσότερο να προστατεύσουμε και την ελευθερία έκφραση. Άρα έχουμε ένα τεράστιο δίλημα να αντιμετωπίσουμε και σε άλλες δύσκολες στιγμές όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια διλήμματα, θα πρέπει να δούμε τι λέει ο νόμος. Και ο νόμος λέει ξεκάθαρα τι είναι απαγορευμένο. Η ρητορική μίσους που μπορεί ε, να προκαλέσει ανοιχτή βία κατά ομάδων ανθρώπων, είτε αυτές είναι μειονότητες, είτε είναι ομοφιλόφιλοι, είτε είναι άνθρωποι με αναπηρία. Είναι κάτι που πρέπει να απαγορευτεί να καταπολεμηθεί με κάθε τρόπο. Και οι πάροχοι επιπρόσεων πληροφορικής εργάζονται, εθελοντικά σε αυτήν την κατεύθυνση, βοηθούν να λύσουμε τα προβλήματα. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά ενώπιον της επιτροπή σας, ότι εκεί ήδη καταλαβαίνω ότι είναι μέρος του προβλήματος και δέχονται ότι θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της λύσης. Εξού και είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν ε, μαζί μας ε, στη σύνταξη αυτού του κώδικα διοντολογίας που θα βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στην Ευρωπαϊκή Νομολογία. Διότι τι βλέπουμε σήμερα, ε, τηρούν πιο πολύ την Αμερικανική νομοθεσία. Πρέπει να επιμείνουμε όμως να τηρηθεί η δική μας νομοθεσία και να γίνουν σεβαστές οι δικές μας αρχές. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να έχω να σας δώσω κάποια θετικά νέα για αυτό τον ε, κώδικα θα υπάρξει δέσμευση υπάρχει να διαγράφουν ε, τέτοια μηνύματα ρητορική μίσους μέσα σε 48 ώρες, μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή που ανακαλύψουν αυτά τα σχόλια. Και υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις. Υπάρχει μια πλήρης δέσμη μέτρων, χωρίς βέβαια, παραλαμβάνω, να θίγεται ελευθερία του λόγου για τη δέσμη μέτρων για την προστασία δεδομένων και για το σχέδιο δράσης. Με την έναρξη, με την έναρξη ισχύω του κανονισμού άρχισε και το έργο μας. Δεν τελείωσε διότι Φυσικά και χαίρομαι που έχουμε αυτό τον κανονισμό, το γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και έχουμε και ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης γιατί θα πρέπει να έχουμε μια ομοιόμορφη προσέγγιση για την αφαρμογή του Γενικού Αυτού Κανονισμού μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων. Γιατί σίγουρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, το βλέπουμε ήδη αυτό. Και πολλές φορές όταν πηγαίνω στις συναντήσεις ε, των ε, ε, ποπτών αυτών για την προστασία των δεδομένων, βλέπω ότι αντιλαμβάνονται ίσως διαφορετικά ορισμένα πράγματα και αυτό μπορεί να οφείλεται στις πολιτισμικές διαφορές που έχουμε. Είναι ένα δεδομένο. Αλλά με τον κανονισμό αυτό θέλουμε ομοιόμορφη δέσμη κανόνων, άρα και ομοιόμορφη εφαρμογή. Ας δούμε τις κυρώσεις. Δεν θα έπρεπε στην Ιταλία, για παράδειγμα, για το ίδιο σφάλμα ή την ίδια ενέργεια να ε, επιβάλλεται μεγαλύτερο πρόσημο στην Ιταλία από ό,τι στην Γαλλία. Θα πρέπει λοιπόν να ε, μαζί με τις αρχές ε, να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουν αυτοί τους εσωτερικούς κανόνες εφαρμογής, αλλά το βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα το χρηματοδοτήσουμε, είναι δημιουργία σαφών κατευθύνσεων της επιχειρήσεις, ώστε όλοι για να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου, ώστε όλοι επαναλαμβάνω, να κατανοούν τους νέους κανόνες και τα νέα καθήκοντα που έχουν. Και ελπίζω να είναι βανάγνωστες και εύληπτες αυτές οι γενικές κατευθύνσεις για τους απλούς πολίτες της Ένωσης, για να δουν ποια είναι τα δικαιώματά τους μέσα σε αυτή την αδέσμη μέτρων και κανόνων. Αυτό είναι λοιπόν το έργο μας για φέτος. Επίσης φέτος θα εκπονήσουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ε, εκπατρισμένους. 18. Για τους ειδικούς, συγγνώμη, experts, όχι expats. Για το privacy shield, την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξει, να εποπτεύει, τι με ρωτήσατε, να βεβαιωθούμε ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις Ρωτήσατε για την εθνική ασφάλεια και τέτοια πράγματα. Φαντάζεστε ότι είχαμε πολύ σκληρές συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Μέχρι πέρσι το καλοκαίρι κυριαρχούσε αυτό το θέμα ε, και ήταν ε, αρκετά πρόθυμοι οι Αμερικανοί εταίροι και φίλοι μας να το συζητήσουν. Κάποια στιγμή καταφέραμε να τα συζητήσουμε και θέλαμε τρία πράγματα καταφέρουμε να τους πείσουν να συζητήσουν. Να δούμε ποιοι είναι οι περιορισμοί ε, των ε, εθνικών αρχών ε, εθνικής ασφάλειας και άλλων υπηρεσιών μέχρι που θα έχουν πρόσβαση. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν εκτίμησε την κατάσταση σε σχέση με τα νέα δεδομένα στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Θέλανε λοιπόν μια σαφή περιγραφή ε, των περιορισμών, πάρα πολύ ε, εκτενή ερμηνεία για το πώς ερμηνεύουν τους νόμους τους, τι ισχύει. Βεβαίως, ακόμα παραμένουν εξαιρέσεις όπου εκείνοι στη δική τους νομοθεσία επιτρέπουν ε, στις υπηρεσίες να συλλέγουν ε, έτσι hidden στοιχεία και μαζικά. Αλλά αυτό πρέπει να ρυθμίζεται για μας την νομοθεσία. Δεν έχουμε ακριβώς ένα φαινόμενο εδώ μαζικού φακελώματος, όπου σωστά επικρίνουν ορισμένοι ότι θα πρέπει να υπάρχει προστασία δεδομένων. Η μαζική συλλογή στοιχείων δεν σημαίνει κατά ανάγκη μαζικό φακέλωμα ή μαζική παρακολούθηση. Υπάρχει το θέμα της ανάγκης και της αναλογικότητας. Αναγκαιότητας καλύτερα και αναλογικότητας γιατί χρησιμοποιούμε εδώ και την ε, φρασεολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ε, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο ε, απολύτως απαραίτητη. Οι Αμερικανοί το χρησιμοποιούν και το επιτρέπουν ακόμα και η πιθανότητα να υπάρχει, όχι η απόλυτη ανάγκη. Ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε απόλυτο έλεγχο των εθνικών αρχών ασφαλείας για το πώς έχουν πρόσβαση στα δικά μας δεδομένα. Ποτέ δεν πρόκειται να το πετύχουμε αυτό, ούτε ε, να έχουμε τη δυνατότητα σε Ευρωπαίο πολίτη να αποζημιώνεται ή να προσφεύγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ούτε στην Ευρώπη. Ποτέ δεν πρόκειται να ελέγχουμε απολύτως τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να το καταλάβουμε ε, είναι μια πραγματικότητα. Για το διαμεσολαβητή είναι και αυτό ένα τμήμα της ιστορίας των διαπραγματεύσεων, διότι για κάποια περίοδο επιμέναμε να έχουμε κάποιον από πλευρά μας που να έχει ε, την έγκριση και ε, τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις διάφορες υποθέσεις όταν ζητούν κάποια στοιχεία και όταν υπάρχουν θεμητοί λόγοι, ας πούμε, αποχρόντες να τα ζητούν. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε εμπλοκή οι διαπραγματεύσεις και ήρθαν οι Αμερικανοί ε, μια ιδέα να ε, θεσπιστεί αυτός ο διαμεσολαβητής που να έχει απόλυτη ανεξαρτησία από οποιασδήποτε αρχές εθνικής ασφαλείας. Προφανώς ε, αυτό είναι καλό και δίκαιο και θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις προσφυγές και όλες τις καταγγελίες των Ευρωπαίων πολιτών και να τις χειρίζεται. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν, ε, δημιούργησαν αυτό το, γραφείο ε, διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εξωτερικό. Τώρα όμως ζητείται από την ευρωπαϊκή πλευρά ε, μια σαφής περιγραφή των αρμοδιοτήτων του κώδικα συμπεριφοράς και διοντολογίας και τι πρόσβαση θα έχουμε εμείς σε αυτές τις πληροφορίες. Εγώ το σέβομαι αυτό γιατί ήθελα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες αλλά ε, και ο χρόνος. Και θα πρέπει να τα συζητήσουμε και τα συζητούμε με τους Αμερικανούς. Δεν έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση. Στόχος μας είναι να φτάσουμε ε, σε μια πιο λεπτομερή περιγραφή αυτών όλων των ε, θεμάτων. Έχω ένα κείμενο που περιγράφει τις αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή που είναι και διαμεσολαβήτρια. Κάπως, με κάποιο τρόπο αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη μου. Δεν ξέρω γιατί κύριοι, ε, ξέρετε είμαι και επίτροπος αρμόδια για θέματα φύλου. Εντάξει, αστείευομαι έτσι. Ωραίο στείο λέει η κυρία Γκόμες, πετυχημένο. Ε, προσπαθώ να έχω ίση μεταχείριση και προσέγγιση. Επάς είναι γυναίκα, η διαμεσολαβήτρια ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, την είδα και προσωπικά στην Ουάσιγκτον. Συναντηθήκαμε και κατανοεί πολύ καλά αυτό που ονομάζουμε εμεί υψηλέ προδιαγραφέ και πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πράγμα που δεν είναι τόσο σύνηθε στι Ηνωμένε Πολιτείε παντού. Εμείς είμαστε έτσι, πρωτοπόροι παγκοσμίω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, να μην σας διαβάσω τώρα τις αρμοδιότητες ε, του διαμεσολαβητή, αλλά πραγματικά προσπαθούμε να ε, λειτουργούμε με τρόπο αποτελεσματικό και ε, μεθοδικό. Έγινε και μια ερώτηση ακόμα για το Privacy Shield από την κυρία Σαρχεντίνη. Αν θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και αν υπάρχει ρήτρα αναστολής. Το συζητούμε και αυτό με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Μετά από τη στάση της Ομάδας Εργασίας 29, για να σας βάλω και στα ενδότερα των υπηρεσιών μας τώρα, κατανοούν πάνω κάτω οι Αμερικανοί εταίροι μας τι ζητούμε από πλευρά του και κατανοούν και τις στάσεις της Ομάδας Εργασίας. the Ε, ε λέω ότι θα ξαναρχίσουν από την αρχή διαπραγματεύσεις, αλλά θα βελτιωθούν ε, τα πράγματα, θα ε, προσαρμοστεί και η απόφαση και οι Αμερικανοί ε, κάπως πρέπει να κινηθούν και αυτοί προς την πλευρά μας, να είναι πιο σαφείς οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του οργάνου αυτού του Δεμεσολαβητού και έχουμε και αυτές τις στάσεις της Επιτροπής 29 για την εφαρμογή. Για τη ρήτρα αναστολής τώρα, ε, αυτό αναφέρεται σαφώς στην ε, απόφαση περί συμμόρφωσης ή καταλληλότητας. Θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό, γιατί αυτό το Privacy Shield δεν είναι απόφαση, ο μηχανισμός είναι. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν δουλεύει καλά, όταν κάποιος που έχει δεσμευτεί να κάνει κάτι δεν το υλοποιεί, ιδιαίτερα οι εταίροι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αναστείλουμε χωρίς διαβούλευση. Μάλλον χωρίς ε, κανένα ενδιασμό ή δισταγμό. Αυτά είναι πεντακάθαρα, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι ε, στη λειτουργία αυτού του μηχανισμού και για να τους εντοπίσουμε αρκετά νωρίς θα έχουμε ετήσια αναθεώρηση και αξιολόγηση. Η πρώτη θα γίνει ε, στα μέσα του 2017 για να αξιολογήσουμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός, πώς συμπεριφέρονται ε, οι διάφοροι φορείς, αν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ε, τι λένε οι ανεξάρτητοι παρατηρητές. Ξέρετε, σε αυτή την αξιολόγηση συμμετέχουν διάφοροι και έχουμε διάφορους διάβλους για να αποκομίσουμε μια πραγματικά ε, αντικειμενική εικόνα για το αν πραγματικά λειτουργεί σωστά αυτός ο μηχανισμός, αν είναι μεγάλη βελτίωση και αν εγγυάται την υψηλή προστασία των Ευρωπαίων. Αυτά για τη ρήτρα αναστολής. Για το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, κάθε φορά που το συζητούμε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης, εγώ λέω το ίδιο δεν πρόκειται να αφήσω να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό τέρας που θα είναι δαπανηρό και άχρηστο. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Και το λέω και τώρα, όπως το έχω πει και πέρυσι, επανειλημμένα, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το αρχικό σώμα, ε, την αρχική ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν πρόκειται να αφήσω να συμβεί. Τα άρθρα 1 έως και 35 ήδη έχουν συμφωνηθεί, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν τα πάντα. Για τις αρμοδιότητες λοιπόν του Γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα πρέπει να έχει πραγματικά τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις και την εξουσία να αρχίσει μια δίωξη ε, να επιστρέφει στα κράτη-μέλη. Ε, θα έχει όμως την προτεραιότητα να αποφασίζει πού θα κινηθεί ε, η έρευνα, η ποινική δίωξη και θα έχει και τη διακριτική ευχαίρεια και τη διαδικασία και την εξουσία λήψη αποφάσεων για να φτάσει το θέμα αυτό σε δικαστήριο, εθνικό δικαστήριο πάντα και οποιαδήποτε περαιτέρω αποδυνάμωση ή ξύλωμα είναι αδύνατο. Θα το πω και τον Ιούνιο ε, και είμαι σε πολύ στενή επαφή και τακτική με την Προεδρία και τις χώρες που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κυκλοφορούν κατά καιρούς διάφορες φήμες και πραγματικά αυτό το συχαίνομαι, γιατί δεν ισχύει ότι ε, διαπραγματευόμαστε σε ενισχυμένη συνεργασία. Καμία σχέση. Δεν ισχύει αυτό καθόλου. Εγώ θέλω όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, αλλά αν δείτε τι λένε οι χώρε, ε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στου καθαρού συνεισφορεί και στου καθαρού αποδέκτε του προπολογισμού. Γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη που παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα από όσα καταβάλουν. Ε, support. Και θα πρέπει να είναι όλοι διατεθειμένοι να υποστηρίζουν ε, την εισαγγελία γιατί είναι ένα ειδικό όργανο, άλλο Eurojust. Εδώ πρόκειται για συγκεκριμένα ζητήματα ε, κακουργημάτων εμπορικά, ε, μάλλον εγκλήματα που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν πολύ θετική η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παραμένει και την εκτιμώ πάρα πολύ. Τα λέω πολύ προσεκτικά <laughs> τώρα όλα αυτά. Παίρνω πολύ ισχυρά μηνύματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός εθνικός σύνδεσμος γιατί ε, το γραφείο του Ευρωπαίου ε, Εισαγγελέα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα εθνικά συμφέροντα άρα να δούμε τι είδους σύνδεσμος θα υπάρχει και το ΦΠΑ θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί ως οικονομικό έγκλημα και να είναι και στις εξουσίες του ε, γραφείου του Ευρωπαίου Σαγγελέα. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά έτσι, συναισθηματική στην έκφραση μου να πω ότι θα αγωνιστούμε και θα παλέψουμε, αλλά θα πρέπει να πείσουμε τους υπουργούς και τους υπουργούς οικονομικών. Φανταστείτε αυτό τι μάχη είναι γιατί οι Υπουργοί Οικονομικών αυτό το θεωρούν ακόμα φορολογικό ζήτημα, αλλά είναι του ποινικού δικαίου ζήτημα η απάτη στο ΦΠΑ. Και γνωρίζω πολύ πολύτως ότι εάν δεν έχουμε, πώς να το πω τώρα, αξιόπιστα στοιχεία, ακριβή για το πόσο χρήματα ε, θα επιστρέψει στο κοινό κουρβανά ε, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ε, δεν θα τους πείσουμε και εγώ δεν θα αφιστώ επιχειρημάτων. Τώρα συλλέγουμε στοιχεία από τα κράτη-μέλη και πιστέψτε με ότι είναι δύσκολο γιατί σε μερικά κράτη-μέλη δεν γίνεται καν διάκριση ανάμεσα ε, στην παραβίαση και την, και την, και ε, την ε, βλάβη στα οικονομικά συμφέροντα του κράτους μέλους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δούμε ε, το πεδίο εφαρμογής, τα όρια, πόσες περιπτώσεις το χρόνο περίπου αναμένουμε να έχουμε, για ποια τάξη μεγέθους μιλούμε, για τι κακουργήματα, για ποια τάξη υποσών. Όλα αυτά εξαρτώνται ε, και θα καθορίσουν ε, και το οργανόγραμμα και το πόσο θα μας κοστίσει αυτή η εισαγγελία. Λοιπόν, έχουμε καλούς λόγους να πιέζουμε τις χώρες, αλλά και για το ΦΠΑ χρειάζεται ακριβώς ε, καλή εκτίμηση για το πόσες υποθέσεις ε, μιλούμε. Το σοβαρό ε, διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα, η απάτη του ΦΠΑ νομίζω θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Από εκεί πέρα βλέπουμε πώς και τι. Έρχομαι στους ανήλικους τώρα implementation of GDPR, I said. On the... Για τους ανηλικούς. Δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο κανόνων και δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να αναλυφθούν για να βοηθηθούν ιδιαίτερα στα ανηλικά. Σε καταστάσεις ε, πολύ δύσκολες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Αυτά λοιπόν τα καθήκοντα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον συνάδελφο που είναι υπεύθυνο για θέματα ασύλου, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι όποτε χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια, θα πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε τα παιδιά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους ανηλίκους ε, σε ό,τι αφορά τα hot spots και σε ό,τι αφορά την αλλαγή λόγω της συμφωνίας με την Τουρκία και σε ό,τι αφορά την συμφωνία με την Τουρκία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα στην Τουρκία πηγαίνουν στους ανήλικους, όχι όλα, αλλά 300.000 αν δεν απατώμε είναι ο αριθμός των παιδιών που δεν έχουν πάει στο σχολείο για χρόνια. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να δαπανηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι και θα πάνε και φυσικά πόροι στους ειδικού οργανισμούς. Σε ό,τι αφορά τη Frontex και τη νέα στρατηγική του 2016 που περιλαμβάνει ιδιαίτερες δράσεις για τα παιδιά σε καταστάσεις τέτοιες μετανάστευσης, δευτερείς γραμμές και ούτω καθεξής πέρα από το σχετικό εγχειρίδιο για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων προκειμένου να εντοπίζουν τα παιδιά σε κίνδυνο. Και το θέμα της κυδαιμονίας των παιδιών σε περιπτώσεις μετανάστευσης, ιδιαίτερα και έτσι ό,τι αφορά την ε, με την κατάσταση των παιδιών σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι ευρύτατο το έγγραφο αυτό, περιλαμβάνει πολλές ε, περιπτώσεις και πληροφορίες και θα πρέπει σύντομα να εφαρμοστεί Να προτείνω, λέει η Πρόεδρο, να περάσουμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων και θα έχετε την ευκαιρία φυσικά να ξαναπάρτε το λόγο για να απαντήσετε στι περαιτέρω ερωτήσει. Ναι, δεν ε, απάντησα όμω για την συμφωνία πλαίσιο. Θα είμαι τώρα πάρα πολύ αυστηρή, λέει η πρόεδρο. Δύο λεπτά, το πολύ. Ο κ. Σκρίπεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γιώργα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας, ε, γιατί μιλήσατε ε, πολλή ώρα και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτά που βλέπουμε ότι περιλαμβάνονται και στο έγγραφό σας. Μιλάτε για τον εξυγχρονισμό των ε, φυλακών, για διάφορα έργα και project. για έργα για την προστασία των πλέον αδύναμων ομάδων, για προγράμματα στις φυλακές και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί πραγματικά ξέρουμε τι γίνεται με την ρίζοσπαθικοποίηση στις ε, φυλακές και ξέρουμε που οδήγησε κιόλας Εξέπλημα χρήματος τώρα τα χρήματα στην Τουρκία, οι πόροι στην Τουρκία που δίνουν στην Τουρκία για την κατάρτιση των παιδιών είναι πραγματικά απαραίτητη και είναι εξαιρετική η δουλειά. Και είναι και μεγάλη δεσμεύση από δική σα πλευρά. Έχω διάφορε ερωτήσει που θα ήθελα να θέσω. Οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση στάζονται υπέρ τη ε, ε, των ίσων ευκαιριών. Και θα πρέπει σίγουρα να επισημάνουμε ότι υπάρχει υποστήριξη των κοινοτήτων ΛΟΑΔ, αλλά γιατί δεν χρησιμοποιείται η ίδια βοήθεια για τις γυναίκες, για τις εγγύους, για τις οικογένειες των αναπήρων, γιατί δεν υποστηρίζονται επαρκώς και αυτοί. Τι αριθμητικά στοιχεία χρησιμοποιείται όταν αποφασίζεται τι γίνεται με τη δαπάνη των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά δεύτερον, πρέπει να ασχολούμαστε πραγματικά με τη μια μικρή περιορισμένη ομάδα ανθρώπων που αλλάζουν διαρκώς ε, φίλο. Ε, δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λόριστεν, ευχαριστώ πολύ γιατί ήρθατε και μας δώσετε πολύ εκτεταμένες απαντήσεις, αλλά μου έχουν μείνει κάποιες απορίες. Ό,τι αφορά τη ρητορική μίσος καταρχάς, είπατε ότι προετοιμάστε ένα κώδικα διοντολογία συμπεριφορά. Μελέτη αντικτύπου, γιατί ξέρετε είναι πολύ ε, μικρή διαχωριστική γραμμή μεταξύ ε, που μπορεί να οδηγήσει και σε λογοκρισία. Αυτές οι δραστηριότητες λοιπόν που θα είναι μια πρωτοβουλία των παρόχων, πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να γίνουν λογοκρισία. Στατιστικά αποδεικνύεται ότι αυτό το μέτρο μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο. Δεύτερη ερώτηση για τα δεδομένα. Είπατε ότι η Frontex εκπονεί τώρα μια νέα στρατηγική που θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων. Πρόσφατα είχαμε εδώ μια μεγάλη συζήτηση για τα δεδομένα με τη Europol και τους λοιπούς. Όλοι αρχίζουν να συλλέγουν δεδομένα και μετά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν κενά σε διάφορες βάσεις δεδομένων. Και δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα, παραδείγματο χάρη. Για τους ε, πρόσφυγες δεν υπάρχει ε, σαφής δομή από πού έρχονται, τι εκπαιδευτικό υποβαθρό έχουν. Ούτε την ηλικία τους δεν γνωρίζουμε. Άρα υπάρχει ένα σχέδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να παρακολουθεί συστηματικά. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για συλλογή προσωπών, δεν για στατιστική παρακολούθηση, στατιστικό έλεγχο της δομής ε, των προσφύγων, των χαρακτηριστικών, του προφίλ τους για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν. Μιλήσατε επίσης για την πρόληψη και αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, μιλήσατε για ίντερνετ και για φυλακέ. Όμως, φυλακές, συγγνώμη. Τι γίνεται όμως με τους καταβλισμούς προσφυγούν και τα hot spot. Και τέλος έρχομαι στη διακίνηση. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση με τη Eurojust ε, καταλήξαμε στο ότι η διακίνηση των ανθρώπων δεν μπορεί να διωχθεί εύκολα. Με αυτό το νέο γραφείο Ευρωπαίου Αγγέλα μπορούμε να περιμένουμε θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κύριε Αγιώτοβα. Ευχαριστώ πολύ. Τρία σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, βέβαια να ευχαριστήσω την Επιτρόπου που ήρθε και ελπίζω να μα δώσει και συγκεκριμένε απαντήσει. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Μιλήσατε διαμακρών για τη μελλοντική στρατηγική και για το, γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Όμω, σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε του, δεν μα είπατε και πολλά. Ούτε για το ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί, η μέθοδο εργασία του. Άρα δεν είναι σαφές ακόμη αυτό. Δεύτερον, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προτείνεται ορισμένα μέτρα και πάλι θέλετε να προβείτε σε αναθεώρηση της οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος. Μα πριν 6 μήνες αναθεωρήθηκε, πολύ πρόσφατα. Επίσης μιλάτε για ένα κώδικα διοντολογίας, συμπεριφοράς, καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Δεν αρκούν αυτά κατ' εμέ. Είμαι στο κοινοβούλιο 7 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια ακούω και ξανακούω ότι ναι, θα υπάρξει συνεργασία και από τους παρόχους ε, του διαδικτύου χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Εγώ όμως θέλω να δω συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Τρίτον, και πολύ συγκεκριμένο και αυτό το ερώτημα, το οποίο αφορά την έκθεση της Σοφίντβελτ με το κρατός δικαίου. Προτίθεστε να προτείνετε ένα νομοθετικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας ε, του δικαστικού συστήματος όλα τα κράτη-μέλη ιδίω ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο. διότι έχω την εντύπωση πως δεν θέλετε και τόσο πολύ να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα για όλους αυτούς τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθηση. Για τη Βουλγαρία-Ρουμανία, για το δικαστικό σώμα κτλ. Πολλά χρήματα δαπανώνται, αλλά χωρί αποτέλεσμα κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλώς ορίσατε, Επίτρε θα είστε τόσο θέματα ίση μεταχείριση και του ε, ΛΟΑΔ. Ήταν αυτό το θέμα τη ε, ίση μεταχείριση ε, θέμα προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την Ολλανδική Προεδρία λάβατε όμω τη σχετική έκθεση Προέδρου την, του Συμβουλίου. Ε, τι περιμένετε λοιπόν, γιατί είχαμε ακούσει ότι πρόκειτο ε, η νομοθεσία για την προσβασιμότητα να επηρεάσει την νομοθεσία σε, για την ίση μεταχείριση. Χρειαζόμαστε τη μεταχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις, ε, τα θέματα ε, ιδιοκτησία ε, μετά από γάμο και σε ό,τι αφορά τα ζευγάρια που είναι, ζουν υποκαταχωρισμένοι σύμβαση εμ, συμβίωσης. Τι ισχύει λοιπόν για τα ζευγάρια ίδιου φίλου, γιατί δεν προβλέπεται τέτοιος ε, γάμος σε όλες ε, τις χώρες. Τι πληροφορίες λοιπόν έχουμε από αυτού. Σε ό,τι αφορά την αύξηση τώρα της ελευθερίας μετακίνησης των οικογενειών ΛΟΑΔ. Τι άλλα σχέδια έχετε, σκόπευετε να διευκολύνετε λοιπόν την μετακίνηση όλων μεταξύ άλλων και της οικογένειας ΛΟΑΔ, γιατί αυτό προαγάγει και τα δικαιώματα των παιδιών. Αν το δούμε από πλευρά των παιδιών, θα ξεκινήσετε λοιπόν μια σχετική πρόταση. Και τι γίνεται με, το... με τα έγγραφα λήξη αρχείου. Και στο σημείο αυτό θα σταματήσω, αν και δεν έχω εξελίσει το χρόνο μου. Μάλιστα. Δεν ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Έχω και εγώ τι δικέ μου ερωτήσει, λέει η πρόεδρο, και μετά. Να, να συνεχίσω στο θέμα των ανηλίκων. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε από την Επιτροπή δεν είναι να κάνει μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε 10.000 αγνοούμενα παιδιά. Συγκεκριμένη δράση χρειαζόμαστε τώρα. Τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά, για να βοηθήσουμε τι ελληνικέ αρχέ που ψάχνουν αυτά τα αγνοούμενα παιδιά τα οποία πλέον εκτίθενται σε ένα σωρό κινδύνους στα, στα των ε, κέντρων αυτών υποδοχής. Τι θα γίνει λοιπόν με τους εισαγγελείς, τι θα γίνει, ποιος είναι ειδικός τελικά με τα παιδιά αυτά, για τους ανήλικους, τους συνοδευτούς. Και μου προκαλεί εντύπωση το τι καθυστερεί την ε, ε, ανάληψη δράσης για την, για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην τελευταία νομοθεσία. Όχι μόνο τα τρομοκρατικά χτυπήματα, αλλά και τα έγγραφα του Παναμά είχαμε προσφάτως. Άρα, το κρίσιμο ζήτημα είναι να αντιμετωπίσουμε φυσικά πρόσωπα να απαγορεύσουμε το σύστημα σύστασης τέτοιων εταιριών. Και πώς το προτείνετε να έχει ένα δικό της τέτοιο σύστημα αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την δέουσα ε, επιμέλεια, σε ό,τι αφορά τα άτομα με πολιτική έκθεση στην Επιτροπή μας είπατε ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα δικό μας σύστημα για να γνωρίζουμε ποιος είναι πολιτική προσωπικότητα εξέχουσα και ποιος όχι. Ευχαριστώ να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις σας για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Γιατί όντω δεν το απάντησε το θέμα αυτό προηγουμένω. Να κατανοήσετε τι κάνουμε. Η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος εγκρίθηκε πρόσφατα και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρω στα κρατημέλη. Την άνοιξη του 2017 θα ολοκληρωθεί. Και υπάρχει μήνυμα προς τα κρατημέλη να ενισχύσουν τις μονάδες για τον έλεγχο του οικονομικού εγκλήματος. Θα πρέπει να έχουν τις, στο σωστό εξοπλισμό για να έχουν και να βρίσκουν τις σωστές πληροφορίες. Και σε ό,τι αφορά τα μητρώα των δικαιούχων ιδιοκτητών. πραγματικών δικαιούχων ε, έχει ήδη εγκριθεί στην αναφερμένη μορφή της οδηγίας. Θέλουμε τώρα λοιπόν να επιταχύνουν τα κράτη-μέλη, να ξεκινήσουν ε, την τήρηση των μητρών αυτών μέχρι τα τέλη του ετού. Δεν μπορώ να σα υποσχεθώ όμω οτιδήποτε, από τα κάτι μέλη εξαρτάται. Η αδυναμία του συστήματος είναι ότι μόνο όσοι έχουν αποδεδεγμένα έναμο συμφέρον μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά και να πάρουν πληροφορίε στα μητρώα αυτά. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, κατέληξα στο λογικό ερώτημα του Μα τι θα γίνει με τους δημοσιογράφους. Με όσους έχουν ε, γενικά τέτοια συμφέροντα. Πώς θα αξιολογηθεί το ένομο συμφέρον τους. Γι' αυτό λοιπόν και στην πρόταση που θα καταθέσω την 1η Ιουνίου, προτείνω να είναι δημόσια τα μέτρα αυτά για να μην χρειάζεται να κρίνουμε το ποιο έχει δικαίωμα και ποιο δεν έχει δικαίωμα να τα συμβουλευτεί. Τώρα, να μιλήσω το, για το τι κάνουμε ήδη για την τροποποίηση της οδηγίας κατά του ξεκλήματος χρήματος. Εξετάζουμε το θέμα των καταπιστευμάτων, των τράστ που δεν ε, χρησιμοποιούνται σε όλα τα κρατημέλη εξίσου. Σε κάποια κρατημέλη δεν υπάρχει η νομική πρόβλεψη αυτή. Υπάρχουν και κάποια κρατημέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως, ε, που όπου αυτό ε, αποτελεί κομμάτι της παράδοσης. Αλλά και πάλι βλέπουμε ε, περιπτώσεις όπου έχει γίνει κατάχρηση των τραστ αυτό για να ξεπλύνεται χρήμα και να φοροδιαφεύγει ο κόσμος. Και αυτό αποτελεί ένα σύνηθες ε, δίλημα να ενοχλούμε τους, ε, τον ειλικρινή και έντιμο πολίτη επειδή υπάρχουν λίγοι ανέντιμοι. Γιατί αποτελεί και κάτι ιδιωτικό αυτό, το τμήμα της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου. Σε κάποιες περιπτώσεις, λοιπόν, ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι περίεργη να δω τι θα έχει ως αποτέλεσμα η μελέτη τύπου. Αλλά κάτι τέτοιο θα χρειαστεί και σε ό,τι αφορά τα τραστ. Στην τελική ανάλυση ενδεχομένω το κράτος μέλος να αποφασίζει αν θα είναι ανοιχτά τα μητρώα αυτά ή όχι. Αυτή η μέση οδό ίσως ισως επικρατησει Τώρα, τι γίνεται με τα έγγραφα του Πάναμα, τα θέματα φορολογική διαφάνειας. Θέλουμε ένα κατάλογο με τις ε, πιο επικίνδυνες, αν θέλετε, χώρες. Και όπως σας είπα, να ενισχύσουμε το ρόλο και τη θέση των ε, υπηρεσιών για τη φορολογική, το φορολογικό έλεγχο. Να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο σε κάθε κράτος μέλος για να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα για τους τραπεζικούς λογαριασμού. Σε κάποια κρατημέλη ήδη έχει πάρει μια κεντρική διάσταση αυτή η δυνατότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα την τρομοκρατία και την πάταξη τη τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εξετάζουμε διάφορα μέτρα, διάφορες λύσεις ε, για τα εικονικά νομίσματα που ήταν ε, ουσιαστικά πέρα από το φάσμα του νόμου. Το βασικό ζήτημα το οποίο συζητάμε, ωστόσο, είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των ανώνυμων προπληρωμένων ε, καρτών. Και εδώ πάλι έχουμε το ίδιο ζήτημα. Ενοχλούμε τον νομοταγή πολίτη ή όχι γιατί ουσιαστικά θα καταργήσουμε την ανώνυμη διάσταση των καρτών αυτών για τις αγορές στο διαδικτύο. Θα ζητάμε από τους καταναλωτές, από τους αγοραστές να δώσουν ένα όνομα, να ταυτοποιήσουν ποιοι είναι και κατά πάσα πιθανότητα θα πέσει και το όριο από 250 σε 150 ευρώ. Αλλά αυτό είναι ακόμη υποσυζήτηση. Αλλά πιστέψτε με, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της οδηγίας για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, πάντα έχω υπόψη μου το θέμα της αναλογικότητας, για να ξέρω μέχρι πού θα πρέπει να φτάσουμε, γιατί αυτό πραγματικά θα σημαίνει ότι θα ε, δυσκολέψουμε τους ε, πολίτες αυτούς στην Ευρώπη, τους νομοταγείς. Από 1η Ιουνίου λοιπόν θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας όταν θα υποβάλουμε τη σχετική προτάση στο ε, Σώμα των Επιτρόπων. Για τα παιδιά τώρα τι κάνουμε ε, για την ασφάλειά τους. Να ε, καταγράφουμε, να ανοιχνεύουμε και να προστατεύουμε τα παιδιά. Το 2016 θα έχουμε μια νέα υποκατηγορία προειδοποίηση στο σύστημα ε, ενημέρωσης ε, και πληροφόρησης για αγνοούμενα ασυνόδευτα ανήλικα. Παιδιά. Ε, τώρα θα μου πείτε, εγώ σας ρώτησα τι θα κάνετε τώρα, όχι την νομοθεσία θα έρθει, αλλά τώρα τι κάνουμε. Λέτε. Βεβαίως θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και να τις εντείνουμε στην καταπολέμηση των διακινητών. κοιτάξτε, βανάκια δεν υπάρχει ούτε κάποιες λύσεις μαγικά Υπάρχουν και κοινέ ομάδες ερευνά, το ακούσαμε, το είπε κάποιος εδώ, είτε στη Eurojust είτε μεταξύ των κρατών μελών και αυτές οι κοινέ διοκτικές ομάδες ε, τα γνωρίζουν. Κάθε φορά που συζητώ με επαγγελματίε του κλάδου μου λένε ότι μπορούν πολύ γρήγορα να έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στη δράση Αλλά η διακίνηση ανθρώπων είναι τόσο κερδοφόρα σε αυτή την κρίση που ανθίσταται σε κάθε δράση που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τώρα βλέπετε κλείνει ο δρόμος των Βαλκανίων και τους έχουν μετατοπίσει προς τα ε, ε, παράλια της Μεσογείου. Δηλαδή είναι και πάρα πολύ ευέλικτη και επίμονη και επιβιώνει αυτός ο κλάδος. Ε. Άρα χρειάζεται ισχυρή πάταξη. Για την ίση μεταχείριση Πραγματικά πιστέψτε με, κυρία Λούνατσεκ, είναι ένα έσχος εδώ. Από το 8 εκρεμίγω, ήρθα το 2014 και κάθε φορά που ανοίγω αυτό το θέμα το ίδιο ακούω. Ότι α, δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για τα, τις κατασκευές, για τα αμαξίδια. Ε, δεν ξέρω ότι είναι πρόβλημα αρμοδιοτήτων. Ακούω διάφορα πράγματα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι στο Συμβουλίο χρειάζεται μοφωνία για αυτό το θέμα θα πρέπει να προχωρήσουμε και πάλι η Ολλανδική Προεδρία υποσχέθηκε ότι θα επιδείξει στένος και πυγμή, κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν μπορώ να σας ε, υποσχεθώ ότι θα εγκριθεί ακόμα ε, η Προεδρία των Κατοχωρών. Εμείς θα πιέσουμε όσο μπορούμε, αλλά πραγματικά νομίζω κάτι κρύβεται πίσω από αυτό, δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει. Για κάποια κράτη-μέλη είναι υπερβολικά λεπτό και ευαίσθητο το θέμα, αλλά θα πρέπει να πιέζουμε και εμείς για να το θέτουμε κάθε φορά επιτάπητος. Είναι πολύ περίεργο. Θυμάμαι σε κάποια συμβούλια, κάποια κράτη-μέλη έλεγαν ότι αυτό το θέμα είναι τόσο σοβαρό και τόσο σημαντικό που δεν θα θέλαμε ποτέ να μπει στην ενισχυμένη συνεργασία. Έτσι, τα ακούμε και αυτά. Δεν λέει αυτό η συντριπτική πλειονότητα, αλλά αν δεν έχουμε ομοφωνία δεν προχωράει. Για το σύμφωνο συμβίωσης, για θέματα γάμου, ιδιοκτησίας, καταχωρημένα ζευγάρια. Είναι δύο νομοθεσίες τώρα, πακέτο θα τις δούμε και θα τις ε, χειριστούμε μας προβλημάτισε. Αλλά η Πολωνία και η Ουγγαρία δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να το δεχτούν και συνεχίσαμε να τα έχουμε σε δύο νομοθετήματα. Παράλληλα, κινούμαστε προς την ενισχυμένη συνεργασία για την έγκριση στο Συμβούλιο τον Ιούνιο κανονικά. Έτσι συμφωνήθηκε η διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι καλό που όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από αυτά τα δύο, έχουν εκφράσει ε, την άποψη ότι δεν θέλουν περαιτέρω καθυστέρηση. Πόσα χρήματα ρωτήσατε επενδύουμε για τις διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού. Δεν το μετράμε έτσι, ότι δίνουμε λίγα λεφτά επειδή είναι λίγοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε μία κατηγορία. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα, αλλά αξίζει ο κάθε άνθρωπος την προσοχή μας και την υποστήριξή μας. Δεν το μετράμε έτσι. Αυτό είναι η ε, ουσία, η κεντρική ιδέα της δημοκρατίας, ότι είμαστε ισχυροί όταν υποστηρίζουμε τις μειονότητες, ανεξαρτήτως αριθμών. Αυτή είναι η ισχύ της δημοκρατίας. Ναι, για τους ΛΟΑΔ, επενδύουμε και για ε, πολλές άλλες αντίστοιχες ε, δράσεις και κατηγορίες. Τώρα προετοιμάζω ένα σχέδιο για μια πολύ σκληρή καμπάνια, εκστρατεία ε, για το 17 που θα καλύψει το φοβερό ζήτημα της βίας κατά των γυναικών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το φαινόμενο στην Ευρώπη. Και κάνουμε ακόμα πολλά περισσότερα που νομίζω ότι πρέπει να γίνουν. To the rights Γιατί θα πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να ε, παρακολουθούμε αυτά τα θέματα συνεχώς. Για τα μετρήσιμα αποτελέσματα, και αυτό που ρώτησε η κυρία Λάουρεστη, για την τεχνολογία της προφορίας. Εγώ ήθελα να έχουμε κάποιους δείκτες στη συνεργασία με τους παρόχους βελτιώνεται η κατάσταση. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι μετρήσιμα. Δεν ξέρουμε πώς αυξομοιώνεται, πώς το λένε αυτό, το φαινόμενο της βίας και της υποδάβλησης του μίσους με, με ε, τέτοιους λόγους μίσου. Πραγματικά εγώ έχω καταβασανίσει τους συναδέλφους μου και τους είπα φέρτε μου δείκτες να μετράμε τέτοια πράγματα και πώς αυτή η δράση έχει αποτελέσματα. Δεν γίνεται αυτό. Βεβαίως παρακολούθηση, έλεγχος και τα λοιπά ε, της κατάστασης είναι εκ των όνων Και κοιτούμε και τις, ε, στρατηγικές, ε, συγγνώμη, τις στατιστικές για τις ποινικέ διώξεις στα κράτη-μέλη, αλλά πώς αλλιώς να το ελέγξουμε. Τι κάνουν οι πάροχοι ίδιοι θα τους ελέγξουμε τι κάνουν, αλλά είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους. Αλλά εμείς έχουμε τον πρώτο λόγο σε αυτό το παιχνίδι, να τους πούμε ε, πού να κατευθυνθούν, να τους καθοδηγήσουμε και με βάση την ομολογία, πού σταματάει η ελευθερία της έκφρασης και τι ε, κόκκινες γραμμές δεν θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτό είναι η δική μας δουλειά, γι' αυτό δείχνουμε τέτοια προσοχή και επενδύουμε πάρα πολύ στην ε, εκπόνηση αυτού του κώδικα δεοντολογίας που δεν έχει να κάνει μόνο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και πώς αυτό ερμηνεύεται ως προς την ελευθερία της έκφρασης. Αυτή η ζώνη είναι αρκετά περίπλοκη και γκρίζα, γιατί άλλη ανοχή ή άλλη επίκαια δείχνουν τα δικαστήρια ανάλογα με τη χώρα. Α, για τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα. Έχουμε διάφορα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση για τα συστήματα αυτά. Τα έκρηση και διάφορα άλλα συστήματα που έχουμε για την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Έχουμε και ενα σύστημα εισόδου-εξόδου που καταγράφει αυτά τα στοιχεία. I must say I uh, Πρέπει να σας πω ότι για αυτή την ερώτηση δεν είμαι πολύ καλά προετοιμασμένη να σας δώσω την απάντηση για όλα τα συστήματα. Πάντως, η γενική μου διεύθυνση και εγώ πάντα φροντίζουμε να είναι δεδομένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα συστήματα. Γιατί αυτό είναι μόνιμο μέλημα και καθήκον μας. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Big, story. Μεγάλη υπόθεση. Ε, πώς προκύπτει η ριζοσπαστικοποίηση είπαμε βασικά είναι στις φυλακές και στο διαδίκτυο. Αυτές είναι οι δύο βασικές πηγές από τις έρευνες που γίνονται, από τις μελέτες. Διαπιστώνει κανείς ότι αυτό δεν αφορά μόνο την ποινική δικαιοσύνη ή τουλάχιστον δεν θα πρέπει να αφορά. Γιατί πρέπει να γίνουν πολλά πολύ νωρίτερα, γιατί άμα φτάσει να γίνει ποινικό, καήκαμε. Αυτό μας λένε και οι πυρογνώμονες, να ψάξουμε τα αίτια. Γιατί ριζοσπαστικοποιούνται οι νέοι. Υπάρχουν λόγοι προσωπικοί, άλλοι οικογενειακοί, από την κοινότητά τους, το περιβάλλον τους, ε, το διαδίκτυο, αν έχουν πρόσβαση, ισχυρή ιδεολογία. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες διαφορετικοί και κάθε ε, ένας από αυτούς τους παράγοντες χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετικά μέτρα. Γι' αυτό είναι το φαινόμενο αυτό τόσο περίπλοκο και τόσο επικίνδυνο παράλληλα. Και αυτό έχει να κάνει και με θεμελιώδη δικαιώματα. Βεβαίως είναι πολύ ευαίσθητο. Αυτά. Τι ώρα είναι. Α, ε, το κράτος δικαίου ε, και ποινική δικαιοσύνη. Το, ο πίνακας επιδόσε αυτό το scoreboard βαθμολόγιο. Να σας πω τι κάνουμε ε, με τη Γενική Συμφωνία Ομπρέλα. Σύμφωνα με το άρθρο 218 κάθετος 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναπόκειται στο Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει απόφαση που να επιτρέπει την υπογραφή της Γενικής Συμφωνίας. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεχώς θα κάνει μια τέτοια πρόταση και θα την δηλαδή θα την εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί αναλόγως. αυτή τη στιγμή υπογραφεί η συμφωνία και με την ε, σύμφωνη γνώμη του, την έγκριση του Κοινοβουλίου θα λάβει απόφαση το Συμβούλιο. Αυτή είναι η διαδικασία και η συγκεκριμένη διατύπωση των όσων κάνουμε τώρα ε, με την δικονομική έννοια, τη, διαδικασία. Ρωτήσατε για ε, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες. Νομίζω ότι προηγουμένως το απάντησε αυτό. Θα πρέπει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρομαι, θα έχει την προτεραιότητα να διώκει και να ε, απαγγέλει κατηγορία, εκτός αν αποφασίσει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να το παραπέμψει σε κράτος μέλος. Θα υπάρχει ένας επικεφαλής ε, εισαγγελέα και μετά τμήματα της εισαγγελία και ε, συνομιλητές στα διάφορα κράτη-μέλη, εντεταλμένοι εισαγγελείς. Όλα αυτά θα γίνονται βάσει της εθνικής ποινική δικονομίας και ποινικού κώδικα, ε, επί της ουσίας δηλαδή σε κάθε κράτος μέλος. Εμείς ερχόμαστε να προσθέσουμε ένα επιπλέον στρώμα πάνω από τα εθνικά, ένα ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ισχυροί χωρίς να θίξουμε ε, το εθνικό δίκαιο. Αν θέλουμε να εναρμονίσουμε το εθνικό ποινικό δίκαιο κάθε χώρας, αν είχαμε τέτοια πρόθεση, ουδέποτε αυτό θα γινόταν πραγματικότητα. Είναι σχεδόν αδύνατο κάτι τέτοιο. Ε, ο Ευρωπαίος εγγελέας δεν θα ε, διώκει ούτε θα ερευνά για θέματα λαθρεμπορίου, οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας κτλ. Το είπα από την αρχή. Εδώ πρόκειται για οικονομικό έγκλημα κατά, κατά των συμφερόντων των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ εξειδικευμένος φορέας. Πώς μετράμε την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας για Όταν ε, μπήκαν οι δύο χώρες αυτές, δεσμεύτηκαν και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ε, benchmarks. Στη Βουλγαρία πήγα πρόσφατα και υπάρχουν τρία-τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουν φέτος. Και, και ο Πρωθυπουργό και οι αρμόδιοι τα θεωρούν εφικτά αυτά. Και εγώ προσωπικά. Εργάζονται πολύ σκληρά για τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα όμως αυτά, όχι μόνο δηλώσεις προθέσεων και την αηφορία και τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων. Ότι η κυβέρνηση να αλλάξει αυτά τα πράγματα θα παραμείνουν και δεν θα καταργηθούν. Για το κράτος δικαίου πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά της Σοφή Ινετβέλτ διότι είναι άχαρο αυτό το θέμα και καθόλου εύκολο το συγκρίνω με αυτό που κάνουμε για το βαθμολόγιο για τη δικαιοσύνη, το scoreboard. Αν δούμε την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη και τη συγκρίνουμε, χρειαζόμαστε ποσοτικούς δείκτες. Δηλαδή, πόσο διαρκεί ε, μία υπόθεση για να εκδικαστεί, πόσες υποθέσεις εκκρεμούν και πόσες υποθέσεις έχει κάθε δικαστής. Μέχρι τώρα ε, είναι καλοί αυτοί οι δείκτες, αλλά από εκεί και πέρα όταν πρόκειται για την ανεξαρτησία, αυτό είναι υποκειμενικό. Δεν μπορείς να το μετρήσεις με κάποιο δείκτη ποσοτικό και πώς θα βρούμε δείκτες από το ευρωβαρόμετρο. Είναι θέμα αίσθησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ε, σε πολλά κράτη-μέλη αυτό είναι άδικο. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τώρα και άλλους δείκτες και άλλα δεδομένα. Και αυτή η παράμετρος της ανεξαρτησίας είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ δύσκολο και καμία φορά και άδικο απέναντι σε κάποια κράτη-μέλη. Από εκεί και πέρα, πώς μετράει κανείς τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Πώς γίνεται αυτό. Εδώ έχει να κάνει με την ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες εξουσίες και τη διάκριση των εξουσιών. Αυτά σας τα λέω από την εμπειρία μου για το πίνακα επιδόσεων της δικαιοσύνης. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, εκτιμώ πολύ τη δουλειά σας κυρία Νίτφελτ. και θα κοιτάξουμε να δούμε ένα τρόπο να συνεργαστούμε. Τώρα, αν χρειάζεται ναι, περισσότερη νομοθεσία, δεν νομίζω. Υπάρχει συνθήκη με μια πάρα πολύ σαφή θεώρηση για το τι εστί κράτος δικαίου και ποιες παράμετροι θα πρέπει να πληρούνται και από τι θα πρέπει να απαρτίζεται. Τώρα ασχολούμαστε με την Πολωνία και προσπαθούμε να το αξιολογήσουμε με τρόπο αντικειμενικό και ευφύ. Ε, με την περίπτωση αυτή ενός κρατου μέλους και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να έχει αντικειμενική αξιολόγηση για ένα κράτος μέλος, έτσι. Και πιστέψτε με, δεν χρησιμοποιούμε καθόλου ποιοτικά κριτήρια, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν, δεν μετερά αυτό το πράγμα με ποιοτικά, με ποσοτικά, συγγνώμη, κριτήρια. Κοιτάμε γενικά την ατμόσφαιρα, το κλίμα, τις τάσεις επικίνδυνες που αναπτύσσονται σε κάποια κράτη-μέλη και θα πρέπει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι και πιο σταθεροί αλλά και πιο ευανάγνωστοι σε αυτά που ζητούμε και αυτά που κατανοούμε εμείς και πώς ορίζουμε το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω και με χαρά να τα ξαναπούμε ε, με μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Επίτροπε, είμαστε ακριβώς στην ώρα μας. Πήγε πολύ καλά τηρήσαμε το πρόγραμμα. Μπορεί αυτό βέβαια να οφείλεται και στο ότι ήταν όντες αρκετοί συνάδελφοι, αλλά έτσι είχατε περισσότερο χρόνο για να μας δώσετε τις δικές σας εξηγήσεις. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και προσβλέπουμε σε μια επόμενη ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Κύριε Γιούροβα, θέλω να σας ευχαριστήσω αξιότιμοι βουλευτές για την δυνατότητα που μου δώσατε να συζητήσω μαζί σας αυτά τα θέματα Δεν μπορώ να σας πω βέβαια ότι είναι ό,τι πιο ευχάριστο για μένα αυτές οι ακροάσεις, αλλά παρόλα αυτά πιστέψτε με ότι προσβλέπω στο μεταξύ μας διάλογο. Φαντάζομαι θα έχουμε στο μέλλον και άλλες ευκαιρίες στην Επιτροπή σας, Πρόεδρος. Τουλάχιστον σας δίνει, πιστεύουμε, αυτή η ανταλλαγή απόψεων μαζί μας περισσότερη δύναμη στη δράση σας στο πρόσωπο της περάσουμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης. Σχέδιο έκθεσης για τη θέσπιση ενωσιακού καινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής. η κυρία Σιλβίγκη Όπως γνωρίζετε, Δεν υπάρχει επί του παρόντος ε, κοινός ενωσιακός κατάλογος ασφαλών χώρων καταγωγή. Κάποιε χώρε έχουν δικού του καταλόγου, αλλά δεν υπάρχει ανταλλαγή, δεν υπάρχουν κοινοί κατάλογοι. Στόχο τη πρόταση τη Κομισιόν λοιπόν είναι η θέσπιση ακριβώ ενό τέτοιου ενωσιακού κοινού καταλόγου βάσει κοινών κριτηρίων, όπω αυτά ορίζονται στην Οδηγία 2013 32 κάθε Ευρωπαϊκή Ένωση για τι κοινέ διαδικασίε, χωρίση ε, ή άρση διεθνού προστασία. Θα δώσω το λόγο καταρχά στην εισηγήτρια εν συνεχεία φυσικά στου Σκιώδης και σε οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο θέλει να λάβει το λόγο. Θα ακούσουμε επίση ε, του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου. Κύριε Κιγιώμη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επανειλημμένω αυτή την πρόταση και εγώ προσωπικά είχα την ε, ευκαιρία να εκφράσω ερωτηματοκά και επιφυλάξει απέναντι σε αυτό το κείμενο οι οποίε επιφυλάξεις, για να σας υπενθυμίσω, αφορούν ε, το κατά πόσο πραγματικά μπορεί να εναρμονίσει κάτι αυτή η πρόταση, γιατί η έγκριση ενό ευρωπαϊκού καταλόγου χωρών ασφαλούς, ε, ασφαλών χωρών καταγωγής δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα οδηγήσει σε πλήρη εναρμόνιση, διότι συνυπάρχει με τους εθνικούς καταλόγους οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Έχω επιφυλάξεις και για την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό των ασφαλών χωρών καταγωγής. Δεν υπάρχει σαφής μεθοδολογία που να προτείνεται μέχρι στιγμή στην πρόταση. Όπως και δεν υπάρχει αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης των 7 χωρών που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον κατάλογο. Έχω επίσης επιφυλάξεις και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης των λόγω καταλόγου διότι δεν είναι σαφής η σχέση αυτού με τους εθνικούς καταλόγους. Ούτε προβλέπεται ένας ευέλικτος, θα ένα επαρκώς ευέλικτος μηχανισμός στη διαδικασία αναστολής. Άρα έχω επιφυλάξεις και σίγουρα άλλοι συνάδελφοι έχουν τις δικές τους. Θα μπορέσουν να τις αναφέρουν στη συνέχεια και μπορεί να αφορούν γενικότερα την έννοια αυτή καθεαυτή της αρχής ασφαλούς χώρας ε, καταγωγής. Τώρα, η προσέγγιση που ακολουθήσαμε, καταρχάς, θελήσαμε και θεωρήσαμε απαραίτητο να υπάρξει ενημέρωση και πληροφόρηση. Πρώτον, να αξιολογήσουμε τις χώρες περιλαμβάνοντας τον κατάλογο. Και δεύτερον, από κοινού με το Συμβούλιο, ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξη Ασύλου ΕΑΖΟ συμπληρωματικέ και θα έλεγα και επικαιροποιημένε πληροφορίε για τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, που αναφέρονται στον κατάλογο. Επίσης αυτό το έργο πληροφόρησης ολοκληρώθηκε αφού επιληφθήκαμε και, μάλλον στραφήκαμε και στον Οργανισμό Θεμελιδών Δικαιωμάτων για να δούμε τι έχει να μας πει σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει αυτός ο κατάλογος στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή, την, σε αυτή τη φάση και το τονίζω, σε αυτή τη φάση αποκλείονται προσωρινά, εξαιρούνται προσωρινά οι χώρες στον κατάλογο από τη συζήτηση για τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο. Περιμένω ε, να λάβω ε, τη συνεισφορά του ΕΑΖΟ για τις ιδεολογικές σκέψεις λοιπόν και τα παρατήματα δεν έχω να πω κάτι αυτή τη στιγμή και το ίδιο ε, αυτή την προσέγγιση θέλω να πω της μερικής εντολής την υιοθετεί και το Συμβούλιο. Οι δύο συνομοθέτες νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει στα άλλα τμήματα του κειμένου και όταν θα έχουμε λάβει τη συνεισφορά του ΕΑΖΟ θα συμπληρώσουμε τη συνεισφορά μας. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι θα περιμένουμε στο δινεκές για την αξιολόγηση των προτινόμενων χωρών. Απλά περιμένουμε πραγματικά ε, επιστροφή που ζήτησε Συμβούλιο και, και Κοινοβούλιο και που απαιτεί και το δικαστήριο. Θέλουμε να υπάρχουν στέρεα θεμέλια για να μπορεί να αξιοποιήσει ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις διατάξεις στο Συμβούλιο. Θέλουμε επίση ενίσχυση τη αρχιτεκτονική ε, του καταλόγου με βάση τέσσερι προτεραιότητε. Σύντομα θα σα τι αναφέρω. Πρώτη προτεραιότητα. Διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκού Καταλόγου και Εθνικών Καταλόγων. Πρέπει να διευκρινιστεί για να έχουν την βέλτιστη δυνατή εναρμόνιση. Θα προτείνω με μεταξύ άλλων διαγραφή των εθνικών καταλόγων εντό προθεσμία τριών ετών και στο μεταξύ σαφεί διαδικασίε για την περίπτωση αναστολή ε, διαγραφή μια χώρα από τον κατάλογο. Πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερη προτεραιότητα. Ενίσχυση τη μεθοδολογία αξιολόγηση των τρίτων χωρών στο πλαίσιο τη διαδικασία ένταξη ή αναθεώρησης του καταλόγου. Αυτό έγκριση συγγνώμη, ή ε, αναθεώρησης του καταλόγου θα πρέπει να υπάρχουν εκθέσεις και επιτόπιες πληροφορίες. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται, δική μας επιθυμία είναι αυτό, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επίσης, αυτή η μεθοδολογία πρέπει να υπαρχουν εκθεσεις και επιτοπιες πληροφοριες και αυτο θα πρεπει να γινεται δικη μας επιθυμια ειναι αυτο απο μη κυβερνητικες οργανωσεις επισης αυτη η μεθοδολογια πρεπει να ενισχυθει και να προβλέπει μια σαφή διαδικασία αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τον κατάλογο. Άρα, θα πρέπει να αιτιολογούνται οι τροποποιήσεις να τεκμηριώνονται με βάση πληροφορίες των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπουμε τη δημιουργία μιας γνωμοδοτικής επιτροπής πληροφόρησης για τις χώρες ασφάλους καταγωγής με μόνιμα μέλη από την ΕΑΖΟ, από την Πατερμοστία του Πρόσφυγε, αλλά θα έχει και μη μόνιμα μέλη, τα οποία θα επιλέγονται με βάση την εμπειρία του για τι τρίτε χώρε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποστολή της Επιτροπής θα ορίζεται σε κάθε στάδιο της ε, διαδικασίας ορισμού ή περαιτέρω κατάρτισης συμπλήρωση του καταλόγου. Για να προλάβω κάποιες παρατηρήσεις, να σας πω ότι όταν προβλέπουν να μπορεί μια γνωμοδοτική επιτροπή να βοηθά στις αξιολογήσεις ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, ίσως ε, μεγαλύτερη γραφειοκρατία, να περιπλέξουμε τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου αυτός ο στόχος μας. Ίσα ίσα, το αντίθετο, θέλουμε να είμαστε πιο επιχειρησιακοί και να ενισχύσουμε αυτή τη ε, διαδικασία και τέτοιου είδους δομές άλλωστε. Δεν είναι κάτι το οποίο εφευρίσκουμε εμείς, αλλά εμπνεόμαστε από το βρετανικό παράδειγμα. Τρίτη προτεραιότητα μηχανισμός αναθεώρησης του καταλόγου που θα είναι πιο γρήγορος και πιο ευέλικτος, διότι ξέρουμε, και θα μπορούσαμε να το δούμε πολύ γρήγορα, ότι μπορεί να υπάρξει μια πολύ ραγδαία αλλαγή ε, στην κατάσταση, ό,τι αφορά δηλαδή ε, την ασφάλεια μιας δεδομένης χώρας. Δεν θα πρέπει να καθυστερούμε πολύ να αντιδράσουμε. Ούτε να κινδυνεύσει να τοποθετηθεί μια χώρα σε ένα κατάλογο που δεν θα έπρεπε να ε, είναι εκεί. Και τέταρτο, η προτεραιότητα να ε, επαναπροσδιορίσουμε το διαδικαστικό πλαίσιο. Έχουμε τι διαδικασίε, την οδηγία για τι διαδικασίε. Η θέσπιση ενό κοινού καταλόγου απαιτεί μια τεκμηριωμένη, αιτιολογημένη ε, ανάλυση. Το είπα ήδη αυτό. Αλλά θα πρέπει επίση να εφαρμόζονται πλήρω οι διατάξει τη οδηγία για τι διαδικασίε και ιδίω οι διαδικαστικέ εγγυήσει. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ισχύει και για άλλου ε, σκιώδει συζητητέ. Τώρα, από νομική πλευρά, ίσω να μην είναι τόσο χρήσιμο να το προσδιορίσουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι αν το κάνουμε, είναι σημαντικό για τη χώρα ασφάλους καταγωγής και η Κομισιόν πρόσφατα δημοσίευσε μια ανακοίνωση όπου προτίθεται λέει να προβεί σε αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας και νομίζω ότι είναι σημαντικό για μια ακόμη φορά να αναφέρουμε αυτό το διαδικαστικό πλαίσιο, το δικονομικό μάλλον πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύω του κανονισμού ζητούμε να υπάρξει έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγηση από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις οικονομικέ εγγύσεις που προβλέπονται στην οδηγία για τις διαδικασίες, σε ό,τι αφορά τους ετούντε από χώρε που είναι εγγεγραμμένες από τον κατάλογο. Σα είπα τα ερωτηματικά, σα μίλησα για την προσέγγιση που έχουμε ακολουθήσει για τις ταξιτές έκθεση, προτεραιότητες επίσης για την ενίσχυση τη αρχιτεκτονικής του κατάλογου τη ανέφερα, Ολοκληρώνοντα λοιπόν αναφέρω ότι με τους Σκιώδη συζητήσαμε μακρόν και θα συζητήσουμε και στη συνέχεια και μια τελευταία λέξη. Μην ε, χάσουμε το στόχο μας με αυτό το κείμενο μην του δώσουμε ένα ρόλο που δεν μπορεί να παίξει. Παραδείγματος χάρη, για, για το στόχο της ομάδας ανθρώπων, ε, να έχουμε υπόψη μας και τους υπηκόους αυτών των κρατών. Πρέπει να τα δούμε ψύχρεμα, ώστε η πρόταση αυτή να μην ε, χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ε, διαφορετικών στόχων. Ούτε να υπερτιμήσουμε τη δυνατότητα αυτής της ε, πρότασης ε, στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης και των συμφωνιών που έχουμε συνάψει. Θα ακούσω πάρα πολύ προσεκτικά τις απόψεις των συναδέλφων σχεδόν και των άλλων συναδέλφων, ελπίζοντας ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ω το δυνατόν πιο γρήγορα με την ολοκλήρωση αυτή τη έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ο λόγος είναι... θα πάει την κυρία που αντικαθιστά τη ο ναι. συγκεκριά. Σας ευχαριστώ και θα παρουσιάσω την ε, τοποθέτηση της κυρίας Ρασιδοντάτη και θα διαβάσω λοιπόν αυτά τα σχόλια που έχει. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιγιόμ για τη δουλειά που έκανε για την έκθεση αυτή. Ακόμα και με την ασυνήθιστη αυτή διαδικασία, με χαρά μου διαπιστώνω ότι επιτέλους προχωράμε στο θέμα αυτό. Αυτό ο Ευρωπαϊκό Κατάλογο των χωρών προέλευση, Ασφαλή, των ασφαλών χωρών προέλευση ήταν ε, η ιδέα του Ζαν claude Γιούγκερ για να αντιμετωπιστούν οι πιέσει οι μεταναστευτικέ στα σύνορά μα. Ακόμα και αν η πρόταση αυτή δεν θα επιλύσει τη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μόνη τη, θα πρέπει να δώσουμε, να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο καλά εργαλεία για να αντιμετωπίσει την μεγάλη εισρωή ετούντων άσυλο. Όπω εξήγησε και η συγγήτρια, θα διαπραγματευτούμε για μια μερική εντολή για το Κοινοβουλίο. Αυτό τι σημαίνει ότι το πιο ευαίσθητο ζήτημα, ο κατάλογος των ασφαλών χωρών προέλευσης θα αναβληθεί και πιο μετά. Σε ό,τι αφορά το κατάλογο αυτό, είμαι βέβαια ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιους ε, σωστούς συμβιβασμούς μεταξύ των πολιτικών ομάδων σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της κυρίας Γκυγιόμ να διευκρινιστεί ε, η εθνική η διαφορά μεταξύ εθνικών καταλόγων ασφαλών χωρών προέλευσης και της ευρωπαϊκής λίστας είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνη. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ο στόχος είναι να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κατάλογος, αν και τα τρία χρόνια μπορεί να είναι πολύ φιλοδοξού ως χρονικό διάστημα. Υπάρχουν διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και Όσο ο ευρωπαϊκό κατάλογο δεν είναι πλήρη, κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να έχει δυνατότητα να, να πάει πιο πέρα. Αλλά φυσικά, μακροπρόθεσμα, στόχο είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Συμφωνώ και την πρόταση τη εισηγητριά να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιείται ο κατάλογο. Όχι μόνο σε καταστάσει εκτάκτου ανάγκη και θα κάνω δικέ μου προτάσει μέσω τροπολογίων. προσβλέπονται στη συζήτηση των θεμάτων αυτών με τους συναδέλφους την επόμενη συνάντηση των σκιωδών. Ελπίζω παρ' όλα αυτά ότι θα μπορέσουμε σύντομα να συζητήσουμε την ε, έκθεση αυτή με πλήρη εντολή, συμπεριλαμβανομένη και του καταλόγου των ασφαλών χωρών, προκειμένου να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν και να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, είναι αδύναμη σε ό,τι αφορά την κρίση τη μεταναστευτική. Ευχαριστώ πολύ από το ECR, ε, ο κ. Χαλάλ. Ευχαριστώ κυρία Αγγίγιο το να υπάρχουν οι κανόνες, ε, σαφείς κανόνες για τα άτομα τα οποία τα χρήζουν διεθνής προστασίας είναι βασική προτεραιότητα για μας. Ο αριθμός των ανθρώπων που επιστρέφονται, που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι βιώσιμος και μειώνει και την ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγεί ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτού που τη χρειάζονται πιο πολύ από όλου. Αν θέλουμε να, να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να μειωθούν οι πιέσει σε κάποια κράτη-μέλη, θα πρέπει να εγκριθούν μέτρα τα οποία θα μειώνουν την γραφειοκρατία και να μην την ενισχύουν. Φοβούμε ότι κάποιε από τι προτάσει που κάνει στην έκθεση τη εισηγήτρια ενδεχομένω να αυξήσουν το γραφειοκρατικό αυτό άχθος και η ομάδα μου συμφωνεί με την εισηγήτρια και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προκειμένου να αξιολογούνται οι χώρε οι οποίε θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι στον κατάλογο, θα πρέπει να υπάρχει ε, να μα δίνονται συμβουλέ από εμπειρογνώμονε. Οι εμπειρογνώμονε αυτέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τη Frontex και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για την δημιουργία ενός ε, επιπλέον ε, συμβουλευτικού σώματος με μεγάλη πολυμορφία απόψεων δεν θα βοηθήσει το σύστημα και δεν θα δημιουργήσει και ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα στις απαιτήσει. Αν σκοπός μας είναι σταδιακά να καταργήσουμε τους εθνικούς καταλόγους, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε περιπτώσεις δηλαδή που δεν μπορούν να επιστρέψουν υπηκόους των χώρων σε, ενώ παλιά το, θα το μπορούσαν. Μπαγκλαντέ, Πακιστάν, Γκάνα, Νιγηρία, Νεγάλη, αυτές οι χώρες θα πρέπει να εξεταστούν ως ενδεχόμενες χώρες ε, για τον κατάλογο αυτό, γιατί οι ετούντες άσυλο από τις χώρες αυτές αναγνωρίζονται σπανίω από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και ο σκοπό μα θα πρέπει να είναι να επιδείξουμε φιλοδοξία, όχι να είμαστε περιοριστικοί προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η πρότασή και τέλο, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για έναν στεναρό μηχανισμό αναθεώρηση. Υποστηρίζω την έκκληση τη εισηγήτρια να γίνεται αναθεώρηση δύο χρόνια. Να γίνει αναθεώρηση δύο χρόνια μετά την έγκριση του μέσου του εργαλείου αυτού. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την χορήγηση άσυλο, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργεί και θα πρέπει να επιλύουμε ενδεχόμενα προβλήματα που θα ανακύπτουν. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα νομοθετικέ αλλαγέ και τροποποίησει. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, καθοδήγηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο τμήμα τη αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να είναι να εκτιμούμε κατά πόσον αυτή η εθνική κατάλογη θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνιμα και τελειωτικά και οριστικά από ένα ευρωπαϊκό κατάλογο. Αυτό ο νέο μηχανισμό δεν θα πρέπει να βάλει σε μειονεκτική θέση τα κρατημέλη σε μια εποχή που ήδη έχουν μεγάλα προβλήματα και αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Να ευχαριστήσω τον εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μαζί τη στις επόμενε μήνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Ντεπρέ για του φιλελεύθερου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως και προλαλήσατε συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω την υποστήριξή μου στην κυρία εισηγήτρια και να τη συγχαρώ για την προσωπική της δέσμευση και στράτευση σε αυτό το θέμα, για τη δουλειά της και για την προθυμία της πάντα να συζητάει με τους σκιώδεις, έτσι ώστε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ φυσικά συμφωνώ με την εισηγήτρια και που προς στιγμή φαίνεται να είναι και εκείνη του Συμβουλίου, να είναι μερική εντολή. Δηλαδή, δεν πρόκειται να αποφαθούμε τώρα εμείς για τον κατάλογο. Ακόμα και αν αρχικά είχα καταλάβει ότι το ενδιαφέρον στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αυτό. Στην αιτιολόγηση της δηλαδή, αυτό ήθελε από τη λίστα αυτή, τον κοινό κατάλογο, να μπορέσουμε να ε, επιταχύνουμε ε, την επεξεργασία και διεκπαιρέωση των αιτήσεων ε, των πολιτών αυτών των χωρών για να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες που κάνουν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι και βέβαιο ότι η συγκήτρια θα ρωτήσει. Ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προσεχώ θα καταθέσει ένα νέο κανονισμό για μια κοινή και ενιαία διαδικασία ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τροποποιώντα ή αντικαθιστώντα τη σημερινή οδηγία για τη διαδικασία ασύλου. Τώρα λοιπόν περί τίνο πρόκειται και τι συζητούμε. Ένα τμήμα του πακέτου των δικονομικών ε, στοιχείων έτσι, για την οδηγία αυτή της διαδικασίας. Και ρωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λέει, εμείς τι δουλειά θα κάνουμε εδώ. Θα κάνει ε, νέα οδηγία η Κομισιόν και απομακρύνει το μιλτής από το μικρόφωνο και δεν τον ακούμε. Από εμά τι περιμένει, θέλει από τώρα να αποφανθούμε ή να περιμένουμε τον κατάλογο. Νομίζω ότι κατάλαβα ότι πολύ γρήγορα θα κάνει μια πρόταση. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα άρθρα και πώς θα τροποποιούνται. Έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγκεκριμένα θέματα λοιπόν για την έκθεση της εισηγήτριας της κυρίας Γιγιόμ. Στην αρχική πρόταση λοιπόν ήταν σαφές ότι ένας από τους στόχους της πρότασης ήταν ο εξής να ε, διεκπεραιώνται πιο γρήγορα κάποια αιτήματα των ε, πολιτών των χωρών του καταλόγου. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται κατάλογος, δεν υφίσταται και στόχος. Αλλά από την άλλη η επιτάχυνση δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα σε όλες τις χώρες, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε εναρμονίσει τις προθεσμίες διεκπαιρέωσης, ούτε τις προθεσμίες προσφυγής, ούτε τις επιπτώσεις. Σε ορισμένες χώρες ε, είναι υποχρεωτικές, σε άλλες όχι. Ε, τι γίνεται τώρα λοιπόν, τι πρόταση θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θίξει αυτό το στοιχείο. Γιατί ε, πρόκειται να φέρει μια ενιαία και μοναδική διαδικασία ασύλου. Για να ξέρουμε και εμείς πώς θα κινηθούμε. Να πω τώρα δύο πράγματα για την ίδια την πρόταση όπως έχει αυτή τη στιγμή. Διαφωνώ λίγο με την εισηγήτρια. Προτείνει να δημιουργηθεί ένα συμβουλευτικό όργανο, το οποίο συμβουλευτικό όργανο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΕΑΣΟ, ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας ΟΗΕ για τις πρόσφυγες και ΜΚΟ. Αυτό κάπως με προβληματίζει. Ο ΕΑΣΟ, το Γραφείο Ασύλου, έχει ακριβώς μεταξύ των βασικών της αποστολών να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γράφει αυτό στην περιγραφή των καθηκόντων της. Και είδα ε, τα απορίσματα και συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνη 21 Απριλίου που ζητάει περισσότερες προφορίες για τις χώρε προέλευση από το γραφείο ΕΑΣΟ για το άσφυρο. Στις 6 Απριλίου σε άλλη ανακοίνωση τα ίδια λένε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την ενίσχυση της εντολής του ΕΑΣΟ έτσι ώστε να γίνει ένας πρωταγωνιστής της εφαρμογής του κοινού δικαιώματος ασύλου και δικαίου. Προσωπικά έχω την αίσθηση να θεωρώ το εξή, ότι αν ξεκινήσει μια ενιαία διαδικασία, ο συνομιλητής κατεξοχήν είναι η Άσο, γι' αυτό δημιουργήθηκε. Όταν κάνει μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δική της δουλειά να έχει κάνει προηγουμένως τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, την ύπατη αρμοστία, τους ΜΚΟ κτλ. Ως συνομιλητής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ νομίζω ότι είναι η ΆΣΟ. Ένας από τους οργανισμούς που δημιουργήθηκαν και συστάθηκαν από την Κομισιόν ακριβώς για αυτό το λόγο. Οπότε τι το θέλουμε το συμβουλευτικό όργανο το άλλο. Έχω πρόβλημα, θα ήθελα να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Ποιον έχεις απέναντι σου συνομιλητή και πώς το οργανώνεις όλο αυτό το θέμα και τη διαβούλευση. Για του εθνικούς καταλόγου, συμφωνώ με την εισηγήτρια αυτή τη στιγμή. Έχουμε κοινέ λίστες και κοινά κριτήρια για να εγγραφούν κάπου σε ένα ευρωπαϊκό κατάλογο κάποιες χώρες. Δεν ε, έχει λόγο ύπαρξη μια εθνική λίστα. Μπορούμε να συζητήσουμε τις προθεσμίες τώρα αν είναι σε δύο, σε τρία χρόνια. Αυτό το συζητώ, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Συμπέρασμα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε λίστα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναδιατύπωση της ε, οδηγίας για τη διαδικασία, θα ήθελα ακριβώς να μας εξηγήσουν ποιο είναι το καθεστώς αυτό που καλούμεθα να δώσουμε και αν θα χρειαστεί και αν χρησιμεύσει σε κάτι, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα έχει άλλα σχέδια και προετοιμάζει άλλα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό και θα ήθελα να καλωσορίσω τη συμπερίληψη ενός συμβουλευτικού σώματος στην, παρακολούθηση των ε, χωρών, των ασφαλών χωρών προέλευσης και θα θέλαμε να δώσουμε ε, μεγαλύτερη υποστήριξη σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση αυτή και φυσικά αν εγκριθεί ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος να ισχύει σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε προσθέκη διαγραφή του καταλόγου και μας ανησυχούν όμως διάφορα ζητήματα. Η μερική εντολή ως ιδέα θεωρούμε ότι αποτελεί μια απόπειρα να διαιρεθεί αυτή η πρόταση στα δύο. Αφενός υπάρχει λοιπόν ε, ε, η ιδέα και αφετέρου έχουμε το περιεχόμενο. Και αυτό λοιπόν ε, αναφέρθηκε. Υπάρχουν ανησυχίες σε ό,τι αφορά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις με της Τουρκίας στον κατάλογο και η χώρα προσπαθεί να διαγράψει αυτό το αμφιλεγόμενο ζήτημα από το θέμα, από το φάκελο, από το ζήτημα αυτό. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο αυτό, ε, τον πανευρωπαϊκό. Δύο ζητήματα έχουμε. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα είναι ότι θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να υπάρχει ίση μεταχείριση και θα πρέπει να υπάρχουν, ε, να ηγετούντες άσυλο τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από το που προέρχονται. Και η δεύτερη ανησυχία έχει να κάνει με την ικανότητα αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τροποποιήσει τις την κατάσταση σε ό,τι αφορά για τις ε, χώρες ε, ασφαλούς προέλευσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα νομικά συστήματα μπορούν και θα έπρεπε να διδρούν πιο γρήγορα από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό λοιπόν τα κρατη θα πρέπει να μπορούν να έχουν ε, τις εθνικές τους λίστες βάσει του κοινωτικού και του διεθνούς δικαίου της σχετικής οδηγίας για τις αιτήσεις για ασυλό. Και γενικά όταν δεν υπάρχουν δηλαδή ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις ένοπλης σύραξης, βασανιστεριών και ούτω καθεξής. Και σε ό,τι αφορά τη συμπεριλήψη της Τουρκίας στον κατάλογο των ε, ασφαλών χωρών, ε, θεωρώ ότι οποιοδήποτε αντικειμενικός παρατηρητής θα συμφωνούσε ότι δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται η Τουρκία. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση της. Εκτιμούμε την ε, σταδιακή προσέγγιση, αν και συμφωνούμε προφανώς με αυτά που είπε η κυρία Άντερσον, με τις ανησυχίες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε με σαφήνεια τα κριτήρια και τη διαδικασία και να μην ε, βιαστούμε από πολιτικής άποψης. Κοιτώντας για παράδειγμα την πρόταση για την Συμβουλευτική Επιτροπή. Είναι σημαντική αυτή η πρόταση, θεωρούμε. Το να υπάρχει ένα τέτοιο σώμα. για να αντισταθμίζεται η πίεση από την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι μας υπενθυμίζει τις βασικές αξίες της Ένωσης σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου. Τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στην, διαδικασία, στην ε, οδηγία της διαδικασίας περιλαμβάνουν και χώρες οι οποίες δεν μπορούν και δεν προτίθενται να δώσουν προστασία στους ετούντες ασύλο. Και μιλώ ως πρόεδρος μιας επιτροπής του Κοινοβουλίου για χώρες που περιλαμβάνουν την το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν και θεωρώ ότι θα είναι ενδιαφέρουσε οι συζητήσει για το πώ εφαρμόζονται όλα αυτά σε, σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα, μα ενδιαφέρει αυτό το θέμα της συμβουλευτική Επιτροπής και συμφωνούμε με τα ερωτήματα που ε, τέθησαν σε, για τον ρόλο των συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε, για παράδειγμα, τη Frontex ως εμπειρογνώμονα. Συμφωνούμε και με ένα ερώτημα που ε, έθεσε η κυρία Ντάτη για τη χρονική περίοδο τριών ετών σε ό,τι αφορά τη μετάβαση από τις εθνικές λίστες σε ευρωπαϊκή λίστα. Και έχουμε κάποιες ερωτήσεις ε, ασφαλώς για την αναθεώρηση της λίστας, γιατί φυσικά μπορεί ταχύτατα να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα προέλευσης και άρα χρειάζεται ένα σύστημα το οποίο να προβλέπει μια, ένα μηχανισμό γρήγορης αντίδρασης στις εξελίξεις. Να συμφωνήσω και με κάτι άλλο που είπε ο κ. Λεπρέ. Πού εντάσσεται αυτό στα πλαίσια των προτινόμενων αλλαγών για το σύστημα ασύλου. Εγώ ήμουν δι... συζητήτρια για την αντιγεία για τις ε, για τις προϋποθέσεις και με απασχολεί αυτό ιδιαίτερως. Αν ρωτιέμαι λοιπόν πώς έχουμε διδαχθεί από τις συζητήσεις εκείνες. Η οδηγία αυτή παρόλα αυτά θα λάβει τη μορφή κανονισμού πλέον, το οποίο φυσικά θα έχει τις συνέπειες του. Άρα πολλά λοιπόν συμβαίνουν στο πλαίσιο αυτό. Πού εντάσσεται λοιπόν αυτή η δουλειά στο πλαίσιο του συστήματος ασύλου. Δεν θα πρέπει να μας ξεπεράσουν τα γεγονότα. Και αν τα κρατημέλη μπορούν να αποφασίζουν από μόνο τους, ε, προφανώς ε, θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Ο κ. Λεπρετών, τελευταίος ομιλητής στη συζήτηση αυτή. Merci, euh, Madame la Présidente, de me donner la... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Πολύ ενδιαφέρουσα την προσωπία Μαγκρέπ συνεδριάζει παράλληλα με την παρούσα συνεδρίαση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την τόσο σημαντική δουλειά που έκανε. Είναι πολλά τα ενδιαφέροντα που μας προτείνει. Ε, η ε, αναβολή της συγκεκριμένης λίστας για τις ασφαλείς χώρες γιατί όχι. Ε, τροπολογία 24 για την επίγουσα διαδικασία που παρακολουθεί λίγο τις κατεξιοδότηση πράξης, πολύ ενδιαφέρον. Απ' την άλλη υπάρχουν τρεις προτάσεις που με προβληματίζουν και έχω πρόβλημα δηλαδή. Η τροπολογία 5 και το δεν το λέω με κακία. Είναι λίγο υποκριτικό όμως αυτό γιατί λέει η ε, κοινή λίστα ε, ασφαλών χωρών δεν έχει ως στόχο τη μείωση ε, των αιτήσεων ασύλου των πολιτών των χωρών αυτών. Μα το αντίθετο, ακριβώς αυτό επιζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ας μην κρυβόμαστε. Τώρα λέμε το αντίθετο, νομίζω δεν βοηθάει τίποτα ούτε την αλήθεια να προοδεύσει. Δεύτερη ε, ανησυχία και παράπονο. Ε, οι τροπολογίες 7 και 25 ζητούν να δημιουργηθεί και άλλο συμβουλευτικό όργανο. Μα και άλλο ένα ακόμα συμβουλευτικό όργανο απλούστευση θέλουμε το συντομότερο. Και ε, οι τροπολογίες 8 και 27 είναι η τρίτη κατηγορία ε, που θέλω να απευθύνω γιατί αυτό είναι βαριά κατάφορη παραβίαση εθνικής κυριαρχίας δεν επιτρέπουν σε χώρες ε, ε, μέλη να θεωρούν εκείνες ασφαλείς χώρες ενώ δεν τις θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουν ένα περιθώριο λιγμών. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να πω και πάλι μπράβο για την έκθεση αυτή. Πρωτού δώσω το λόγο στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα από πλευρά μου. Είτε μιλάμε για ευρωπαϊκές λίστες, είτε για εθνικούς καταλόγους. Μήπως βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των ασφαλών χωρών. Αυτό θα πρέπει να το εξετάζουμε ασφαλώς κατά περίπτωση, ανά Γιατί ένα ανθρωπο από το Πακιστάν μπορεί να βρίσκεται σε μια σαφέστατη κατάσταση που να χρήζει ασύλου παρά το γεγονός ότι το Πακιστάν δεν θεωρείται χώρα ασφαλούς προέλευσης. Και το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία. Αν πρόκειται για Τούρκο Κούρδο, για παράδειγμα, ή αν πρόκειται για δημοσιογράφο ενδεχομένω από την Τουρκία. Μήπω λοιπόν βρισκόμαστε σε μια οξύμορη κατάσταση σε ό,τι αφορά το διεθνέ δίκαιο και τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Νίλσον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Uh, δύο βασικές παρατηρήσεις από πλευράς μας. Πρώτα απ' όλα, Είμαστε ευνοϊκώς διακείμενοι στο πνεύμα των τροπολογιών που θέλουν να, uh, να διευκρινίσουν τη συνύπαρξη των εθνικών καταβλών με το μελλοντικό ενωσιακό διάλογο και να δούμε επίσης πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ε, σε μια εναρμόνιση, αν θέλετε, ευρωπαϊκή της αρχής της ασφαλούς χώρας καταγωγής. Αυτές οι τροπολογίες, λοιπόν, ε, μπορούμε να τις δεχθούμε. Κάποιες επιφυλάξεις, όμως, για τη δημιουργία αυτού του νέου γνωμοτικού οργάνου, του νέου συμβουλευτικού οργάνου. Ε, συμφωνώ και εγώ με ορισμένα σχόλια ότι έχουμε την ΕΑΖΟ που υποτίθεται πρέπει να υποστηρίζει όλους τους θεσμούς και φορείς ε, σε ό,τι αφορά την πολιτική ασύλου και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα αρκεί. Και έρχομαι και στην πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν που αναφέρθηκε από ορισμένου. Μεταξύ άλλων βλέπουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το ρόλο της ΕΑΖΟ και πώς μπορούμε να κάνουμε πιο σαφή την εντολή της σε ό,τι αφορά την παροχή συμβουλών προς τα κράτη-μέλη και κυρίως ε, προς ε, τις διάφορες οργανώσεις. Μια κοινή ανάλυση που θα μπορούσε να είναι βάση για μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, σε σχέση με τη συμπερίληψη χωρών στον κοινό κατάλογο. Όπως ανακοινώνουμε επίσης, θα υπάρξει και αλλαγή, τροποποίηση του, της οδηγίας για τις διαδικασίες για να γίνει συγκεκριμένα κανονισμός. Ζητώ την κατανόησή σας, αλλά σήμερα δεν είμαι σε θέση να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Ωστόσο, θεωρώ ότι η πρόταση που έχουμε σήμερα επιτάπητος και την οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα βράχι πρόθεσμο μέτρο που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν ε, την ε, σοβούσα κρίση, αλλά μέσω και μάκρο πρόθεσμα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε το συνολικό πλαίσιο. Και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και την ε, περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών που μπορεί να συμπεριλάβει και την οδηγία για τις διαδικασίες ό,τι αφορά τις ασφαλείς χώρες καταγωγής. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Το θέμα είναι ε, ο χρονισμός. Έχουμε κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα και έπειτα έχουμε και την μέσο μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο εκπρόσωπος της Προεδρίας ή εκπρόσωπος του Συμβουλίου Θέλω να λάβει το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια γιατί στην έκθεσή της λαμβάνει υπόψη ε, τις συνομιλίες που είχαμε πριν από αρκετούς μήνες ε, όταν και είχαμε συμφωνήσει για αυτή τη μερική εντολή σε ό,τι αφορά ορισμένα τμήματα του κειμένου, περιμένοντας ε, και τη συνεισφορά ε, των δύο οργανώσεων, ΕΑΖΟ και Οργανισμού Θεμελιωτών Δικαιωμάτων. Θα περιμένουμε τις ε, πληροφορίες από την ΕΑΖΟ, έχουν λάβει το σχετικό αίτημα. Τώρα, το Συμβούλιο συζήτησε διαμακρών αυτή την πρόταση. Έχει καταλήξει συμφωνία για μια συμβιβαστική πρόταση. Πήραμε διαπραγματευτική εντολή από την Κορεπέρ. Επί της ουσίας τώρα. Δύο σημεία θέλω να τονίσω. Τα οποία συζητούμε στο Συμβούλιο. Το πρώτο. Διάρκεια και επιπτώσεις αναστολής. Της περίοδου αναστολής. Μιας τρίτης χώρας από τον ενωσιακό κατάλογο άρθρο 2 ή 3. Δεν ήταν σαφές όταν δηλαδή έχουμε την εξή περίπτωση. Είναι μια χώρα στον ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών, αλλά αν αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα που απαιτεί την αφαίρεσή της από αυτόν τον κατάλογο, η Κομισιόν μπορεί να προτείνει να ανασταλεί η συμπερίληψή τη, η εγγραφή τη στο κατάλογο. Αυτό είναι μια γκρίζα, μια φαία ζώνη, γιατί δεν μπορεί να μπει η χώρα σε έναν εθνικό κατάλογο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή τη χώρα ούτε και η αρχή της ασφαλούς χώρας προέλευση, ή καταγωγή Το Συμβούλιο για να αποφύγουμε αυτή την γκρίζα ζώνη, ακριβώς και για τους λόγους που αναφέρατε προηγουμένως και εσείς και άλλοι, ότι δηλαδή πραγματικότητα επιτόπου μπορεί να αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε κάνει προτάσεις ως Συμβούλιο και καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική πρόταση. Δηλαδή να είναι έξι μήνες το πολύ αυτή η περίοδος αναστολής και να μην έχει και τόσες μεγάλε δυνατότητε η Κομισιόν να παρατείνει αυτή την περίοδο πέραν το εξαμήνου. Τι περιορίζουμε αυτέ τι δυνατότητε. Δεύτερον, ανάγκη διευκρίνηση στη σχέση μεταξύ εθνικού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγή και του ενωσιακού. Ιδίω όταν μια χώρα έχει αφαιρεθεί από τον ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευση. Εδώ η Προεδρία μα βρέθηκε αντιμέτωπη με τα δύο άκρα. Απ' τη μία αν θα μπορεί να βετάρει η Κομισιόν ε, τη συμπερίληψη μιας χώρας σε έναν εθνικό κατάλογο αφού έχει ε, σβηστεί από, έναν, από τον ενωσιακό ή να αφήσει τις χώρες ε, να διατηρούν στον εθνικό τους κατάλογο μια χώρα που έχει αφαιρεθεί από τον νοσιακό, που δεν είναι και τόσο ευκταίο αυτό ως δεύτερη επιλογή. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία να περιορίσουμε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής την εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορεί να ασκήσει βέτο για τη συμπερίληψη μιας χώρας σε ένα εθνικό κατάλογο αφού έχει η ίδια χώρα αφαιρεθεί από τον νοσιακό κατάλογο. Εδώ ε, σταματώ. Ζητώ συγγνώμη αν ήμουν λίγο γενικόλογος Το κείμενο είναι πολύ πιο σαφές. Περιλαμβάνονται προθεσμίες, χρονοδιαγράμματα στο κείμενο, πολύ συγκεκριμένα αναφέρονται όλα. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι το Συμβούλιο προσβλέπει σε μια επικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι σκόπιμα αγνοεί την ερώτησή μου σε ό,τι αφορά το κατά πόσο συνάδει αυτό με το διεθνέ δίκαιο, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το δίκαιο, την ε, συνθήκη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ε, προσφύγων. Να δώσω το λόγο στην κυρία τη σε που θέλει να απαντήσει. Θα είμαι σύντομη, γιατί πολλά ακούσαμε ήδη και νομίζω ότι η συζήτηση ήταν αρκετά εκτεταμένη. Τρία ζητήματα θέλω να επισημάνω. Ο κύριος από το Συμβούλιο είπε μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ακριβής και σε κάποιες άλλες λιγότερο. Το θέμα όμως είναι να υπάρχει μία ε, ρευστότητα στις εξηγήσει για το πώς ε, λειτουργεί το σύστημα κατάρτισης, διαγραφής ε, σε ό,τι αφορά τον κατάλογο αυτό για να είναι σαφή τα πράγματα, να μην υπάρχουν θέσεις, και δυνατότητες ερμηνείας για την Συμβουλευτική Επιτροπή. Είπα εκ των προτέρων ότι περίμενα σχόλια σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό άχθος που θα σήμαινε. Και περίμενα και τα σχόλια και από τη Βρετανία, καταλαβαίνω τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσουμε και εκεί να δείξουμε μια ευελιξία. Και για το κομμάτι αυτό θα πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτο η ΑΖΟ να είναι νόμιμος συνομιλητής σε ό,τι αφορά τέτοιες ε, προσεγγίσεις. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες για άλλες, από άλλες αυτικές γωνίες. Δεν χρειάζεται να καταστήσουμε μια επιτροπή με 25 άτομα. και σε ό,τι αφορά τις εξελίξει εξελίξεις επιτόπου σε περίπτωση μιας χώρας, για παράδειγμα, και όταν μια χώρα καθίσεται ασφαλής, είναι αρκετό να έχουμε μια-δύο παραπάνω απόψεις που θα επιβεβαιώσουν αυτή την τοποθετήση. Και το τελευταίο ζήτημα, το οποίο έδειξε η κυρία Άντερσον, πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά να γίνει μεγάλος όγκος δουλειά προκειμένου να αποφευχθεί να μην είναι ε, διαδικαστική αυτή, αυτό το σύστημα, διεκπαιρεωτική για τις ροές από χώρα σε χώρα, γιατί θα μπορούσε, ελοχεύτως ο κίνδυνος. Άρα θα πρέπει να μην περιοριστούμε στην ε, τρέχουσα λίστα, θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά αυτή η αρχή σε περιπτώσεις όπου ο κατάλογος αυτός θα ε, είναι μακροπρόθεσμο. Σα ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για τα σχόλια που κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναπληρώσω το σημείο αυτό τη ημερησίας διδάξης. Ε, Προθεσμία είναι για την κατάσταση τροπολογιών 13 Μαου το μεσημέρι. Και νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει και τη σημερινή μα συνεδρίαση. Να σα υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 9 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 στο Στρασβούργο. Μετά θα έχουμε στις 23 και 24 Μαΐου συναντήσεις συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και λίγη έτσι η συνεδρίαση.